Okay, friends, you are warmly welcome to our meeting. Καλώς ορίσατε στη συνεδρίασή μας. Σημείο 1, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δεχτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ανακοινώσεις της Προέδρου στο σημείο 2. Καταρχάς, υπάρχει πλήρες γλωσσικό καθεστώς με την εξαίρεση των κρατικών. Και για αύριο θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι το πρωί Η κυρία Μωρίν Σαρτιέ έχει 20 ε, προσκεκλημένους από την περιφέρειά της για να παρακολουθήσουν τις συνεδρίες της Επιτροπής από τις 9 μέχρι τις 10.30. Σημείο 3. Ενημερωτικά θα γίνει μια έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Απασχόλησης στις 24 Μαΐου. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα εξή. Θα είναι εδώ ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης για το διαρθρωμένο διάλογο και η Επίτροπος Τάισεν επίσης για την πρόταση για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας όπως ζήτησαν οι συντονιστές στις 15 Μαρτίου. θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και μετά θα γίνει ψηφοφορία για το διαρθρωμένο διάλογο και ένα εργαστήριο για την ε, ε, αρχή εργασίας ε, το οποίο οργανώνει το Τμήμα Πολιτικής. Παρακαλώ λοιπόν να είστε εδώ όσο το δυνατόν περισσότεροι. Τώρα, έγκριση των πρακτικών, αν δεν υπάρχουν στάσεις, εγκρίνουμε τα πρακτικά 27 Μαρτίου και περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση, προβλήματα στην αγορά εργασίας και στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Ο στόχος αυτής της συνεδρίασης είναι να συζητήσουμε τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης οικονομίας εν γέννη και κυρίως ε, στην αγορά εργασίας. Υπάρχει μεγάλος βαθμός αβεβαιότητας όσον αφορά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Υπάρχουν ανησυχίες, ελπίδες ένα αμάλγαμα και των δύο και γνωρίζουμε από ένα μια πολύ γνωστή εργασία, η οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές, ε, η οποία δηλώνει ότι ε, το 47% των αμερικανικών θέσεων εργασίας κατά πάσα πιθανότητα θα αυτοματοποιηθούν στην επόμενη δεκαετία, στις επόμενες δύο δεκαετίες. Ε, άλλες μελέτες βέβαια εκτιμούν ότι θα δει το πολύ ένα 10%. Ε, το 47% με το 10% είναι μεγάλη διαφορά βεβαίως. Τώρα, ε, Μαθαίνουμε επίσης ότι ε, θέσεις ε, μέσης, ε, μέσων δεξιοτήτων ε, μειώνονται, αλλά και η υψηλή δεξιότητα θέσεις εργασίας και οι χαμηλή δεξιότητα θέσεις εργασίας επεκτείνονται, αλλά υπάρχουν οι πλατφόρμες, η οικονομία η γη οικονομία και οι εργαζόμενοι θα έχουν, δεν θα έχουν τόσο ωφέλη όσα έχουν οι εργαζόμενοι τώρα, όπως για παράδειγμα άδεια ε, γονική ή ε, αδιασθενείας. Και όλες αυτές οι τάσεις φυσικά θα επηρεάσουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και έχουμε ένα πάνελ. Θα ξεκινήσουμε με μια παρουσίαση της ε, ΣΤΟΑ μία μελέτη για τον αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας και την κοινωνική οικονομία. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Μπέρναρ Τάξ. καταρχάς, ο οποίος θα μας κάνει μια πρώτη εισαγωγή και παρουσίαση της μελέτης της ΣΤΟΑ, αλλά δεν έχει έρθει. Είναι από αυτούς που αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω της απεργίας ε, της Brussels Airlines σήμερα. Ε, προτείνω λοιπόν να δώσουμε το λόγο στους τρεις επιρρογνώμονες πρώτα Μπορείτε να μιλήσετε λοιπόν για 10 λεπτά περίπου καθένας και μετά ελπίζουμε στο μεταξύ να έρθει ο κύριος Ντάξ, ο οποίος είναι καθοδόν. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Σάμουελ Έγκμπλον, ο οποίος είναι Διευθυντής Πολιτικής και πρώην ε, επικεφαλής ε, νομικός σύμβουλος στην ε, TCO, την Σουηδική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Εργαζομένων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και την Επιτροπή σας ε, για την ευγενική πρόσκληση εδώ και ε, για να σας παρουσιάσω τις θέσεις του οργανισμού μας. Ο TCO, ο, η Σουηδική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών ε, Εργαζομένων, έχουμε 4 εκατομμύρια εργαζομένους ε, σε διοικητικές θέσεις ε, και στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Είμαστε μία από τις 10 μεγαλύτερες ε, συνομοσπονδίες στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και είμαστε και από αυτές που αυξάνονται πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, οι νέε τεχνολογίες επηρεάζουν την αγορά εργασίας με δύο τρόπους. Πρώτον, αποτελούν μοχλό διαρθρωτικών αλλαγών και δεύτερον, δίνουν και τη δυνατότητα νέων τρόπων οργάνωσης εργασίας. Και θα διαρθρώσω και την παρέμβασή μου βάσει αυτών των δύο θεμάτων. Αν αποφύγουμε τις πιο δυστοπικές και τις πιο τοπικές ε, ε, προβλέψεις, οι προβλέψεις για τις συνέπειες της ψηφιοποίησης στην αγορά εργασίας συνοψίζονται ως εξής κάποιες θέσεις εργασίας θα χαθούν, κάποιες θέσεις εργασίας ε, θα προκύψουν και οι περισσότερες θα αλλάξουν. Και νομίζω ότι αυτό συνοψίζει και τη μελέτη της ΤΟΑ που θα ακούσουμε αργότερα. Η ταχύτητα των αλλαγών θα είναι διαφορετική μεταξύ των διαφόρων τομέων στις διάφορες χώρες και ε, επίσης και μεταξύ των επιχειρήσεων όταν εξετάζουμε την ψηφιοποίηση δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ποτέ βεβαίως ότι ακόμα κι αν ε, υπάρχει ε, μια πολύ ισχυρή δύναμη που είναι οι τεχνολογικές αλλαγές, οι αποφάσεις ε, σε πολιτικό επίπεδο θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Σε επιχειρηματικό επίπεδο, γρήγορη και λογική προσαρμογή σε τεχνολογικές αλλαγές θα είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αν δούμε το δημόσιο τομέα, ισχύει το ίδιο ακριβώς και η τεχνολογία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες ε, που ε, χρειαζόμαστε και ε, νομίζω ότι το αυτό ισχύει και για τον τρίτο τομέα. Κάτι άλλο στο οποίο συμφωνούν πολλοί εμπειρογνώμονε είναι ότι οι δεξιότητε και η ικανότητα να αποκτήσει κανεί δεξιότητε θα είναι πολύ σημαντικέ. Η ποιότητα του παραδοσιακού εκπαιδευτικού συστήματο από την προσχολική ηλικία μέχρι το πανεπιστήμιο είναι πολύ σημαντική, αλλά επίση θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επιμέλεια στη διάρκεια της ε, ε, εργασιακής ζωής και για αυτούς που μπορεί να χάσουν τη δουλειά του ε, τη δουλειά τους λόγω αλλαγής ή για αυτούς που χρειάζονται εκπαίδευση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές σε ένα συγκεκριμένο τομέα επάγγελμα. Σε μια έρευνα που είναι πολύ σημαντική για την σουηδική αγορά εργασία, βλέπουμε ότι 4 στου 10 εργαζομένου πιστεύουν ότι δεν λαμβάνουν αρκετή μετεκπαίδευση στη δουλειά του για να σταθούν και στο επίπεδο των αλλαγών και αυτοί που ανησυχούν περισσότερο είναι οι μεσήλικες, όχι οι νεότεροι ή μεγαλύτερες ηλικίες έργα. Επίσης αυτοί που έχουν υψηλές δεξιότητες και άτομοι, άτομα με μόνιμες θέσει εργασίας που ανησυχούν... Ε, συγγνώμη, ε, ε με συμβάσεις εργασία ανησυχούν περισσότερο από αυτού που έχουν μόνιμες θέσει εργασία. Επίση θα ήθελα να τονίσω και πόσο σημαντικά είναι να υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας ε, και μια ενεργό αγορά εργασία για να μπορέσουν να μετριάσουν τι αρνητικέ συνέπειε ε, για του αυτού που χάνουν τι θέσει εργασία του, αλλά και να διευκολύνουν και τι τεχνολογικέ αλλαγέ. Αν θέλει οι άνθρωποι να εναγκαλίσουν τι αλλαγέ, πρέπει να του παρέχει και ασφάλεια. Τώρα, η αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών ε, σημαίνει ότι υπάρχουν πολλέ δυνατότητε για τι συλλογικέ διαπραγματεύσει και τι διαβουλεύσει μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Ενημέρωση και διαβούλευση με του εργαζομένου πριν από την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο να γίνει περισσότερο αποδεκτό, αλλά να υπάρχει και καλύτερη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων. Οι συλλογικέ συμβάσει μπορούν επίση να βοηθήσουν ώστε να εξασφαλίσουμε κατάλληλη αναβάθμιση των εργαζομένων όταν αλλάζουν οι θέσει εργασία και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότε να έχουν δικαιώματα αλλά και ευθύνη. Τρίτον, ε, συλλογικέ συμβάσει εργασία σε τομεακό επίπεδο μπορεί να ε, χρησιμοποιηθούν για διμερεί ή τριμερεί οργανώσει ε, που βοηθούν του εργαζομένου που χάνουν τι εργασίε του. Στην τελευταία πρόβλεψη, ο, ΩΣΑ, αναφέρθηκε στα Συμβούλια Ασφαλείας ε, το Σουηδίας ε, και είπε ότι είναι πολύ καλό παράδειγμα. Ελπίζω να το ακολουθήσουν και άλλοι στα πλαίσια των ε, εργασιακών σχέσεων. Οι νέε τεχνολογίε επίση δίνουν τη δυνατότητα για νέου τρόπου οργάνωση εργασία. Η τεχνολογία τη πληροφορική διευκολύνει το συντονισμό τη εργασία που γίνεται εντό και εκτό των φυσικών και νομικών ορίων της παραδοσιακής επιχείρησης. Αυτό επιτρέπει στους εργαζομένους να έχουν ένα μικρότερο εργατικό δυναμικό μονίμων εργαζομένων και να το συμπληρώνουν ε, με συμβάσεις εργασίας, με αυτοαπασχολούμενους και οι άλλοι εργαζόμενοι μπορεί να πάνε πέραν αυτού και να έχουν και ένα επιχειρηματικό μοντέλο το οποίο να βασίζεται σε άτυπες ε, μορφές εργασίας για όλες τους τις ανάγκες. Η ψηφιοποίηση λοιπόν είναι μοχλός προς την κατεύθυνση ε, συντομότερων, πιο ε, περιστασιακών εργασιακών σχέσεων και ένα θέμα το οποίο έχει λάβει μεγάλη προσοχή είναι οι λεγόμενες θέσεις εργασίας πλατφόρμας που σχετίζονται με επιχειρήσεις όπως η Uber, η Fondora, η Task και το Amazon Mechanical Turk. Επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία ε, εργασιών ε, κατά, αναλόγως της ζήτησης ε, έχει λίγη σχέση με την Ήμπε και τη Φοντόρα. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτής των εργασιών είναι από γυναίκες και γίνεται σε παραδοσιακές επιχειρήσεις, για παράδειγμα στη λιανο, λιανική πώληση, στα εστιατόρια και στη παροχή φροντίδας. Σε αυτούς τους τομείς μπορεί να καλείται κάποιο εργασία ή να ακυρώνεται κάποια προγραμματισμένη εργασία που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη ροή των ε, πελατών, και εκεί μπορούμε να έχουμε μεγάλες, ε, ε, μεγάλες πλειονότητες που εργάζονται με μερική απασχόληση ή με συμβάσεις καθώς επίσης και ε, να υπάρχει διαμοιρασμός ε, σε βάρδιες, ε, να δουλεύει κάποιος σε αναμονή ή να έχει και συμβάσει μηδενικών ωρών εργασίας. Επίσης ε, όλα αυτά καθοδηγούνται από την τεχνολογία. Υπάρχουν συστήματα βελτιστοποίησης εργατικού δυναμικών που επιτρέπει στα καταστήματα, στα εστιατόρια και σε παρόχους ε, υπηρεσιών υγείας να αναλύσουν τις ροές των πελατών και να προσαρμόσουν αναλόγως και τα προγράμματα. Ε, εφαρμογές επίσης έξυπνων τηλικών νεφώνων ή απλώς μηνύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλέσει κάποιους εργαζόμενους. Εδώ έχουμε για παράδειγμα τεχνολογικές επιχειρήσεις ε, όπως η Κρόνος, η Infor, η Ceridian, ε, ο ιδιοκτήτης του Dayforce, η Geneson και πολλές άλλες οι οποίες δεν έχετε ακούσει ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι οι κακοί, αλλά απλώς σας ενημερώνω ότι υπάρχουν οικονομίες που είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που, ε, με τον τρόπο που τις βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε τεχνολογικό επίπεδο. Τέλος, έρχομαι σε απαντήσει από πλευρά πολιτική αυτέ τι αλλαγέ στην οργάνωση τη εργασία. Πρώτον, πιστεύω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή του κείμενου κανονισμού για τι νέε μορφέ εργασία. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε ισότιμους όρου εργασία για όλε τι επιχειρήσει που προσφέρουν υπηρεσίε ταξί, μεταφορών και παράδοση. Ε, το να θεωρεί κάποιο ότι είναι πλατφόρμα ή τεχνολογική επιχείρηση δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγει την νομοθεσία που πρέπει να τηρήσουν οι ανταγωνιστέ σου. Βεβαίω θα πρέπει να γίνει προσαρμογή τη νομοθεσία για να επιτρέπει και αυτέ τι νέε τεχνολογίε. Δεν θα πρέπει πρέπει να παρακολύεται η καινοτομία σε καμία περίπτωση. Δεύτερον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευελιξία ε, που υπάρχει στις διάφορες κατηγορίες του εργατικού δικαίου. Πριν σκεφτούμε την εισαγωγή νέων κατηγοριών εργασίας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές που έχουμε. Η έννοια του εργαζομένου ε, έχει αλλάξει ε, την τελευταία τον τελευταίο αιώνα και έχει αποδείξει όμως ότι μπορεί να προσαρμοστεί στις αλλαγές. Και έτσι δεν θα πρέπει να υπάρχουν κλειστοί ορισμοί, ιδιαίτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που ε, ε, είναι και ο λόγος για τον οποίο ε, η δική μου οργάνωση είναι αντίθετο στο συγκεκριμένο σκέλος της οδηγίας για τις γραπτές δηλώσεις. Τέλος, θα πρέπει να μην εισάγουμε νέες τρίτες κατηγορίες σε κράτη-μέλη στα οποία δεν υπάρχουν. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή και τμήματων του εργατικού δικαίου, όπου χρειάζεται για τους αυτοαποσχολούμενους. Ε, για παράδειγμα, αν δούμε τους κανονισμούς για την επαγγελματική ασφάλεια και την υγεία στον χώρο της εργασίας θα μπορούσαν να επεκταθεί στους αυτοαπασχολούμενους ε, που λαμβάνουν οδηγίες και έχουν στενό συντονισμό με επιχειρήσεις πελάτες αλλά χωρίς να είναι εργαζόμενοι της επιχείρησης. Πρέπει επίσης να προσαρμόσουμε τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για να καλύψουν και τις ανάγκες αυτών των εργαζομένων που δουλεύουν κατόπιν ετήματος. Ε, παραδοσιακά αυτά τα συστήματα έχουν ε, κάποιον ο οποίος έχει μία μόνιμη θέση εργασίας ή μία σύμβαση εργασίας με σταθερό εισόδημα. Και δεν καλύπτει αυτούς τους εργαζομένους ε, που είναι αυτοαποσχολούμενοι ή που συνδυάζουν την εργασία ως εργαζόμενοι και αυτοαποσχολούμενοι. Πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθούν αυτές οι κατηγορίες και να προσαρμοστούν τα συστήματα. Σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξουν οι απαιτήσει προσόντων, να αλλάξουν οι κανόνες για τη συνεχή επιλεξιμότητα, ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζονται τα επιδόματα, επιδόματα στην ασφάλιση ανεργίας, ε, τα επιδόματα ασθενείας και τη γονική άδεια για να υπάρχει κατάλληλη προστασία για εργαζομένους που έχουν ε, σύντομα ε, συμβάσεις εργασίας, είναι αυτοαποσχολούμενοι και ή αυτούς που συνδυάζουν εργαζόμενο και αυτοαποσχολούμενο. Τέλος, για τα συνδικάτα. Πρέπει όπως πάντα να οργανωθούμε και για να γίνει αυτό πρέπει να μπορούμε να έχουμε και κάποια συνάφεια με το αντικείμενο. Οι εργαζόμενοι που έχει τρεις διαφορετικούς εργοδότες ε, μπορεί να έχουν μια προσφορά η οποία να αξίζει να συμμετέχει κάποιο στο συνδικάτο. Το, το ίδιο ισχύει και για τους συμβούλους ε, πληροφορικής που είναι αυτοαποσχολούμενοι. Επίσης θα πρέπει να παρέχουμε απτά ωφέλη ακόμα και σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα συλλογική διαπραγμάτευσης. Πρέπει να παρέχουμε συμβουλές για το πώς μπορεί να συμμετέχει κανείς σε αυτό το νέο τοπίο της γκίγκ οικονομίας με τον καλύτερο τρόπο, να τονίσουμε πώς μπορούμε να υπάρχει εξασφάλιση για αυτούς που δεν καλύπτονται από πολιτικές ε, τις οποίες ε, ε, εφαρμόζει ο εργοδότης και αυτός είναι ένας τρόπος να ενισχύσουμε και τα μέλη στην οικονομία αυτή Όσον αφορά την ανάγκη που αναφέρθηκε ήδη να διατηρήσουμε και να αναβοθμίσουμε τις δεξιότητες, τα συνδικάτα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο μέσω παροχή ε, μαθημάτων ε, και ε, να παρέχονται αυτά τα, τα μαθήματα είτε δωρεάν είτε με πολύ χαμηλό κόστος. Και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να συμβάλλουμε στην αποτελεσματική εφαρμογή θα πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να οργανώσουμε τα μέλη μας και να μην υπάρχουν πρακτικά ή νομικά προσκόμματα στην οργάνωση αυτή. Νομίζω τελείωσε ο χρόνος μου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και πολύ ευχαριστώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας αργότερα. Ευχαριστώ. Thank you. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Θα έλεγα να περάσουμε κατευθείαν στο δεύτερο μιλτή και μετά να προχωρήσουμε στις ε, ερωταπαντήσεις. Θα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Ντάξ. Ε, είχα υπόψη να μιλήσετε αργότερα, αλλά αν θέλετε μπορείτε να μιλήσετε τώρα, να μας παρουσιάσετε τη μελέτη της ΣΤΟΑ, γιατί κατ' ουσίαν έτσι θα, ξεκίνησε, θα ξεκινούσε η συζήτηση. Έχετε λοιπόν το λόγο για 10 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που με καλέσατε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για να σας παρουσιάσω κάποια αποτελέσματα της μελέτης. Ζητώ συγγνώμη, αλλά ξέρετε καθυστέρησε η πτήση μου Βέβαια ο συνάδελφός μου κάλυψε αυτό το κενό και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας έκανε μία μελέτη για την ΣΤΟΑ, για τις νέες τεχνολογίες, ε, πώς οι νέες τεχνολογίες θα επηρεάσουν την αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι γνωρίζουμε και είναι προφανές ε, ότι ζούμε σε μια νέα εποχή όπου πλέον έχουμε νέες τεχνολογίες. Βεβαίω αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι αλλάζει η οργάνωση εργασίας, η απασχόληση, το επίπεδο της απασχόλησης στην οικονομία. Αν θέλετε ένα νέο αφήγημα, ε, απλά για να αναφέρω κάποιες ε, νέες τεχνολογίες, ε, έχουμε την, το ψηφιακό εργοστάσιο, την ψηφιακή παραγωγή, ε, το 3D, την εκτύπωση σε 3D. Ε, αυτό είναι επίσης κάτι πολύ καινούριο που έχει πάρα πολλές επιπτώσεις σε αυτά είναι απαραίτητα που χρειαζόμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Έχουμε ε, την αλγοριθμική λήψη αποφάσεων, την τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που σχετίζονται με το λογισμικό και με το πώς μπορεί κανείς να λάβει καλύτερα αποφάσεις με τη βοήθεια της ε, σύγχρονης τεχνολογίας. Έχουμε ε, ρομπότ, έχουμε ε, οχήματα χωρίς οδηγό, αυτόνομα και βεβαίως έχουμε και κάποιες καινοτομίες στον τομέα των ψηφιακών ρυθμίσεων, γιατί έχουμε τα bitcoin και τις ε, τεχνολογίες blockchain. Δεν είναι μία μόνο τεχνολογία, είναι μία σειρά από νέες τεχνολογίες. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται για όλους είναι ε, ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των νέων μορφών τεχνολογίας στην απασχόληση. Και νομίζω ότι για να είμαι ειλικρινής, ξέρετε, δεν ξέρω ποιες είναι οι επιπτώσεις, δεν μπορώ να πω. Η συζήτηση που γίνεται ε, μπορεί να ψηστεί ως εξής. Δεν έχουμε ένα αφήγημα, αλλά δύο αφηγήματα. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα αυτά θα έχουν ε, τεράστιες επιπτώσεις, αλλά δεν ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση. Θα έχουμε ευτυχές τέλος ή ε, θα είναι κάτι που θα πάει τελείως στραβά. Σήμερα δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιο είναι το πιο σωστό από τα δύο αφηγήματα. Επιτρέψτε μου όμως να σας παρουσιάσω αυτά τα δύο αφηγήματα με βάση αυτά που υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Εκείνο λοιπόν που είναι κοινό και για τα δύο αφηγήματα είναι ότι οι μηχανές ή αν θέλετε γενικότερα η τεχνολογία θα αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε. Την καθημερινή δουλειά, τη δουλειά ρουτίνας, αλλά επίσης και τη δουλειά γραφείου. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν πολλές πιθανότητες όλα αυτά να αυτοματοποιηθούν λόγω της τεχνητής ε, νοημοσύνης, λόγω των ρομπότ και πολλών άλλων συναφών πραγμάτων. Αυτό λοιπόν ε, που μπορούμε να περιμένουμε είναι όμως ότι θα υπάρξουν και νέες μορφές εργασίες, νέες ευκαιρίες ε, για ανθρώπους να μπορούν να κερδίζουν τα προστοζή από τελείως ε, διαφορετικό τρόπο εργασίας ε, ή θα είναι δραστηριότητες που δεν θα είναι δραστηριότητες ρουτίνας και θα ε, εναπόξουν ανθρώπους να εργαστούν σε αυτό το νέο πλαίσιο. Σκεφτείτε τι γίνεται με τις τράπεζες. Οι τράπεζες, ναι, πράγματι έχουν εισαγάγει τη νέα τεχνολογία, αλλά τελικά απλά άλλαξαν, επανεκπαίδευσαν το προσωπικό τους και πέρασαν από θέματα ρουτίνας σε θέματα μη ρουτίνας, όπως ε, παροχή συμβουλών στους πελάτες, ε, ε, σχέση, συζήτηση με τον πελάτη. Αν θέλετε, αυτό είναι ένα ευτυχές τέλος και κατά κάποιον τρόπο, αν θέλετε, επίσης το θα οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγικότητα, σε βελτίωση των εισοδημάτων, σε μια νέα μορφή οικονομικής ανάπτυξης ε, που θα ε, δρομολογηθεί από τη νέα τεχνολογία. Ορισμένα επαγγέλματα δεν θα εξαφανιστούν, απλά θα αλλάξουν. Ίσως κάποια πράγματα να εξαφανιστούν, αλλά αρκετά επαγγέλματα θα παραμείνουν και απλά θα αλλάξουν μορφή και περιεχόμενο. Τι θα γίνει όμως αν όλα αυτά πάνε στραβά. Σας είπα προηγουμένως ότι οι μηχανές μπορούν να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους. Ε, ισχύει αυτό σε μεγάλο βαθμό, σε διοικητικές εργασίες, σε χειρονακτικές εργασίες, αλλά πάντα υπάρχει ελπίδα ότι θα υπάρξουν νέα επαγγέλματα, νέες θέσεις απασχόλησης ε, για ανθρώπους οι οποίοι θα εξοικειωθούν με αυτές τις ε, νέες διεργασίες. Ορισμένοι πιστεύουν ότι αυτό πια δεν γίνεται γιατί οι μηχανές είναι καλύτερες σε όλους τους τομείς ε, και πολλοί πιστεύουν ότι θα παραμείνουν πολύ λίγα επαγγέλματα και απλά θα προκύψουν πολλά και καινούργια. Αυτό όμως είναι το κακό σενάριο, γιατί σημαίνει ότι η ανεργία θα αυξηθεί, πολλοί άνθρωποι θα ε, παραμένουν σε επαγγέλματα που δεν μπορούν να αυτοματοποιηθεί και έτσι αναγκαστικά θα συρρυκνωθούν οι μισθοί σε αυτά τα επαγγέλματα. Θα υπάρξει μεγαλύτερη ανισότητα και διχασμός. Και βεβαίως ε, θα ασκηθεί και επίση τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ε, γιατί τα συστήματα κοινωνική ασφάλιση βασίζονται σε ε, υψηλά ποσοστά απασχόλησης. Αυτά είναι ε, τα δύο σενάρια. Το ένα είναι αποδεκτό, το άλλο όχι, αλλά τελικά ποιο είναι το πιο πιθανό να συμβεί. Αυτό το ερώτημα ετέθη στη μελέτη μας. Τι μπορούμε να μάθουμε από την εμπειρία μας με την τεχνολογική αλλαγή και πώς μπορούμε αυτά να τα εφαρμόσουμε σήμερα. Θέλω να πω το εξή. Αυτή η, ένταση ανάμεσα στι νέε τεχνολογίε, οι οποίε καταστρέφουν επαγγέλματα, όμω δημιουργούν και νέα επαγγέλματα, αυτό δεν είναι καινούριο. Αυτό υπάρχει από τη βιομηχανική επανάσταση. Υπάρχει πάντα αυτό ο αγώνα ανάμεσα στην καταστροφή και τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων. Και όπω σα είπα, κατά το παρελθόν πάντα επικρατούσε η δημιουργία νέων επαγγελμάτων. Και γι' αυτό και εγώ είμαι αισιόδοξο και πρέπει να, είναι, να ισχύει για όλους, να είναι όλοι αισιόδοξοι. Πιστεύω ότι το αίσιο τέλος είναι πολύ πιο πιθανό να συμβεί από ένα δυσάρεστο τέλος. Βεβαίω υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν, να ληφθούν υπόψη. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Διότι έχουμε το διαδίκτυο, το οποίο σήμερα είναι πολύ πιο διαδεδομένο από ό,τι ήταν κατά το παρελθόν. Ε, Παραδείγματο χάρη είναι το ηλεκτρικό ρεύμα η τεχνολογία με βάση τον ατμό. Αυτές ήταν εφευρέσεις ε, που μπορούν να συγκριθούν λιγάκι σήμερα με το διαδίκτυο αυτού του επίπεδου. Η ε, τεχνολογία, αν, η πληροφορική και επικοινωνία, οι τεχνολογίες σε αυτούς τους κλάδους ε, έχουν ακόμα ένα τεράστιο δυναμικό. Ως εκ τούτου αυτές οι τεχνολογίες ε, μπορούν να κάνουν μετά από δύο-τρία χρόνια πράγματα που ούτε καν να τα σκεφτούμε δεν μπορούμε σήμερα. Και βεβαίως ε, έχουμε και το εξής φαινόμενο ότι πάρα πολλά πράγματα που είναι ψηφιακά μπορούν να αναπαραχθούν με πολύ περιορισμένο κόστος. Αυτό είναι κάτι που διαχωρίζει την ε, ψηφιακή οικονομία από όλες τις άλλες ε, μορφές τεχνολογικής ανάπτυξης που είχαμε κατά το παρελθόν. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ σε θέματα πολιτικής και τελειώνω την ομιλία μου. Πιστεύω ότι αυτά που πρέπει να γίνουν είναι προφανή και όλοι θα συμφωνήσουν ότι οφείλουμε να επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση. Είναι αλήθεια ότι η δουλειά ρουτίνας ε, κατά το μέλλον θα περιοριστεί και νομίζω ότι πρέπει τα εκπαιδευτικά συστήματα να τα επαναπροσαρμόσουμε σε διαπροσωπική επαφή. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη. Βεβαίως και πρέπει να επενδύσουμε και στις υποδομές και νομίζω ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό, αλλά δυστυχώς πολλοί το αγνοούν ότι πρέπει να κάνουμε και περισσότερα για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Γιατί αν δούμε τις ε, νέες τεχνολογίες, ε, πρόσφατα υπήρξε μία μελέτη για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δούμε λοιπόν αυτές τις ε, νέες τεχνολογίες, νομίζω ότι η Ευρώπη είναι πολύ καλή στο επιστημονικό κομμάτι, όμως υπάρχει έλλειψη επιχειρηματικότητας. Θα ήταν λοιπόν πολύ καλύτερα αυτές τις τεχνολογίες να τις εφαρμόσουμε στην αγορά, γιατί μέχρι τώρα απλά επικρατούν οι μεγάλες εταιρείε, εταιρείε από την Κίνα. Θα ήταν καλύτερο να επικρατούν οι ευρωπαϊκές εταιρείε στην Ευρώπη. Και με αυτά τα λόγια θα ήθελα να κλείσω την ομιλία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντάξ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον καθηγητή Βαλέριο Ντεστέφανο καθηγητής στο Ινστιτούτο Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Λέβεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επιτροπή σας για αυτή την ε, πρόσκληση. Ακούσαμε δύο παρουσιάσεις επί των ποσοτικών πτυχών σε ό,τι αφορά την επιρροή που θα ασκήσουν οι νέες τεχνολογίες ε, ε, στην αγορά εργασία, αλλά εγώ είμαι νομικός, δεν μπορώ να σας πω τόσο λοιπόν για τα ποιοτικά, ποσοτικά στοιχεία όσο για τα ποιοτικά. Γιατί ε, συχνά αμελούμε αυτό το ζήτημα στη γενικότερη συζήτηση για τις νέες τεχνολογίες και την αυτοματοποίηση θα ήθελα πρώτα να, πω, να σταθώ στο βασικό μου μήνυμα σήμερα εδώ. Πρώτον, απαιτείται διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες ε, και πώς χρησιμοποιούνται και οι νέοι αλγόριθμοι για, την, για να δοθεί κατεύθυνση στην αγορά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένας σωστός κοινωνικός διάλογος για την αλγοριθμική διαχείριση ε, του, ε, εργατικού δυναμικού. Το δεύτερο που ακούσαμε και από τον προηγούμενο μιλητή είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε από τις ετικέτες της απασχόλησης ε, και της ε, παροχής ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να περιορίζουμε λοιπόν τέτοια δικαιώματα όπως είναι το δικαίωμα στην συμμετοχή σε συνδικάτα και το καθεξής μόνο για τους υπαλλήλους. Πρέπει να τα διευρύνουμε αυτά τα δικαιώματα. Και πρέπει να εξετάσουμε την απασχόληση ως μια ευέλικτη έννοια που σε ορισμένε περιπτώσεις θα πρέπει να ε, αναδιοργανωθεί για να μην εξαιρεί τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων. Όταν μιλούμε για την ψηφιοποίηση, πολλές φορές αναφερόμαστε στην οικονομία πλατφόρμας ε, που αφορά ε, εργασία που μπορεί να γίνει και στο διαδίκτυο και εκτός, ε, αλλά συνδέεται με νέες τεχνολογίες όπως είναι η Uber και το καθεξής. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι συχνά ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι εργαζόμενοι που εργάζονται μέσω πλατφόρμας, ιδίως ό,τι αφορά ε, τους οικιακούς βοηθούς και όσους παρέχουν φροντίδα, που πολύ συχνά τους ε, ξεχνάμε. Είναι λοιπόν παραμελημένη αυτή η κλάδη. Πολύ συχνά όταν έχουν να κάνουμε με εργασία πλατφόρμας, ε, όλοι αυτοί θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι και έτσι δεν έχουν πρόσβαση σε ε, εργασιακή προστασία, βασικό μισθό, ε, συλλογική διαπραγμάτευση και κοινωνική προστασία, κοινωνικής ασφάλισης μάλλον. Σε ορισμένε περιπτώσεις έχουμε και που ε, που μέσω τη πλατφόρμας έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασία Σε άλλε περιπτώσει. Ε, είναι εικονική και μόνο η αυτοαπασχόληση. Γιατί σε ό,τι αφορά την ε, παροχή της ε, εργασίας, παρακολουθείτε με τα ψηφιακά συστήματα, ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας, ο τρόπος και το και εμείς ως πελάτες μπορούμε να αξιολογήσουμε την εργασία τους. Αυτό σημαίνει ότι μέσω αλγορίθμων ασκείται και πειθαρχία, αν θέλετε, προς τους ε, εργαζομένους, αν το επίπεδο παροχής υπηρεσιών ή το χρονικό πλαίσιο δεν ήταν ε, αρκετά ικανοποιητικό, ε, μπορούν να ασκηθούν πειθαρχικά μέτρα ή ακόμα και να αποκλειστεί ο εργαζόμενος από την πλατφόρμα. Όμως δεν έχει σχέση με την πρόσβασή τους στην πλατφόρμα. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι μορφές εργασίας ε, αποκλίνουν από την πραγματική και αυθεντική όπως την γνωρίζουμε εργασία. Στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο βλέπουμε ότι οι εργαζόμενοι σε πολλές ε, περιπτώσεις ε, στρέφονται στα δικαστήρια και ζητούν να καταχωριστούν ως εργαζόμενοι. Σε ορισμένε περιπτώσεις τα έχουν καταφέρει, σε άλλε όχι. Σε πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις και στην Ιταλία και στη Γαλλία είδαμε ότι αξιώνουν την ε, ταξινόμησή τους υπό τους ε, υπαλλήλους, υπό το καθεστώς του υπαλλήλου του εργαζομένου ε, και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχει μια εικονική ευελιξία του χρόνου εργασίας. Τι σημαίνει αυτό. Θεωρητικά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν πότε και αν θα εργαστούν και μέσα στην εβδομάδα και μέσα στην ημέρα τους. Πρώτον, θα πω ότι αυτή η ευελιξία είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο ε, εξαίρεσής τους από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Γιατί υπάρχουν άλλες τέτοιες αρχές. Αν δεν μπορεί κάποιος να αποφασίσει και να επιλέξει τις χρεώσεις του, ε, τον τρόπο που θα υλοποιήσει ε, και θα φέρει σπέρα στο καθήκον του και το χρόνο που θα του πάρει αυτό, ε, ουσιαστικά δεν μπορεί κανείς να εξαιρέσει κάποιον από τα συστήματα κοινωνικής προστασίας μόνο και μόνο λόγω του στοιχείου που προανέφερα. Ιδίως ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία και, τη δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε εάν η υποτιθέμενη αυτή ευελιξία υφίσταται. Σε πολλές περιπτώσεις δεν ξέρουμε πώς οι αλγόριθμοι ε, κρίνουν ένα ευέλικτο χρονοδιάγραμμα. Αν κανείς δεν είναι ε, διαθέσιμος συνεχώς, μπορεί ε, να τιμωρείται από την πλατφόρμα και να δώσει, να δώσει δηλαδή, η πλατφόρμα περισσότερη δουλειά σε άλλους που είναι διαθέσιμοι πιο συχνά. Ουσιαστικά λοιπόν δεν γνωρίζουμε κατά πόσο συμβαίνει αυτό γιατί τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για να αξιολογήσουν ε, τις επιδόσεις ε, και να κατανείμουν το φόρτο εργασίας στο μέλλον δεν δημοσιεύονται. Και αυτό έχει να κάνει και με το θέμα της διαφάνειας στους αλγορίθμους ε, σε επίπεδο διοίκησης και διαφάνεια ε, των ε, συστημάτων αξιολόγηση. Αυτό είναι πολύ ευρύτερο λοιπόν από την ε, οικονομία της πλατφόρμα. Όλο ένα και περισσότερο χρησιμοποιούμε αλγορίθμους, τέτοιε πλατφόρμε και άλλα τέτοια συστήματα για να δούμε ποιου θα πρέπει να προσλάβουμε, ποιου να προαγάγουμε και ποιου να απολύσουμε. Και τώρα χρησιμοποιούνται αυτά τα μέσα για την μέτρηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας όμως δεν τα γνωρίζουμε αυτά τα κριτήρια συγκεκριμένα και εγώ θεωρώ ότι χρειαζόμαστε διαφάνεια. Και ο πιο αξιόπιστο τρόπο για να γίνει αυτό είναι η ύπαρξη κοινωνικού διαλόγου και συλλογική διαπραγμάτευση επί των κριτηρίων που αξιοποιούν οι πλατφόρμες και οι ε, εργοδότε σε πιο συμβατικό επίπεδο για την αξιολόγηση των εργοζομένων. Η συλλογική διαπραγμάτευση είναι ο πλέον κατάλληλο και ευέλικτο τρόπο για να γίνει αυτό χωρίς να διοχετευτεί όλο αυτό σε νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι πολύ πιο δύσκολο να αλλάξουν. Είναι πιο ευέλικτο μέσω λοιπόν η συλλογική διαπραγμάτευση. Προκειμένου ε, να διασφαλίσουμε ότι θα διανοματίσει αυτό το ρόλο η συλλογική διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πάμε πέρα του ε, παραδοσιακού πεδίου εφαρμογή τη συλλογική διαπραγμάτευση. Δεν πρέπει λοιπόν να αφορά μόνο του παραδοσιακού ε, εργαζομένους υπαλλήλους, αλλά και τους αυταπασχολούμενους. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν νομικά προσκόμματα γι' αυτό. Οι αυταπασχολούμενοι λοιπόν να περιοριστούν από την... και να μην τους επιτραπεί να συμμετάσχουν στη συλλογική διαπραγμάτευση, γιατί αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ε, ε, εικονική ρύθμιση των τιμών, price fixing, το οποίο απαγορεύεται από το δίκαιο ανταγωνισμού. Ε, πρέπει λοιπόν να βρεθούν λύσεις ε, για να υπερβούμε τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες. Και τέλος, επειδή δεν μου μείνει πολύς χρόνος, θα πρέπει να εξετάσουμε και τα κριτήρια προσδιορισμού της ε, σχέσης εργασίας κριτήριο όπως η συνεχής διάθεση ενός εργαζομένου προς τον εργοδότη ε, θα πρέπει να λαμβάνει μικρότερη σημασία στο μέλλον. Ιδίω εάν στο μέλλον οι εργοδότες έχουν μια μεγάλη δεξαμενή ε, εργαζομένων που θα μπορούν να κινητοποιούν ανα πάσα στιγμή με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Η δυνατότητά τους να επιλέξουν αν θα εργαστούν ή όχι και πότε ε, και το αν υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει μικρότερη σημασία αν υπάρχουν άλλοι δείκτες που μας ε, δείχνουν ότι υπάρχουν παραδοσιακές σχέσεις ε, απασχόλησης και υπαγωγής. Επομένως, οι τεχνολογικές εξελίξεις θα πρέπει να κινηθούν προς όφελος της κοινωνίας και όχι το αντίθετο. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον επόμενο μιλητή, τον Δ. Γέλλιντ Βίσ Κίρσεν, αντιπρόεδρο του IBAGEI. E Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε το λόγο. Ε, ήμουν συντάκτρια μιας μελέτης ε, του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Απασχόλησης για αυτό το ζήτημα πέρυσι αλλά γενικά είμαι νομικός σε ζητήματα εργατικού δικαίου ε, και τα πρόσφατα σχόλιά μου θα περιοριστούν ακριβώς στα νομικά ζητήματα. Τα βασικά ευρήματα της μελέτης ήταν τα εξή. Πρώτον, είδαμε ότι η ψηφιοποίηση αφορά και τους εργάτες ε, της χειρονεκτικής εργασίας και ε, τους υπαλλήλους γιατί κάποιοι έχουν την δυνατότητα ότι όλοι, έχουν την εντύπωση ότι όλα αυτά αφορούν τη βιομηχανία και τον παραγωγικό κλάδο. Ενώ το 80-90% των εργαζομένων στην Ευρώπη εργάζονται στον κλάδο των υπηρεσιών. Δεύτερον, από τη μελέτη προκύπτει ότι θα υπάρξουν νέες ε, επιχειρηματικές δομές, νέες μορφές απασχόλησης και αύξηση των αυταπασχολουμένων. Τρίτον, η μελέτη έδειξε ότι ενδεχομένως να υπάρχει κίνδυνος μαζικής ανεργίας και καθώς αναφερθήκατε σε μια προηγούμενη μελέτη του 2015 που έλεγε ότι το 47% των ε, ε, θέσεων εργασίας στην αμερικανική αγορά θα εξαλειφθεί. Υπάρχουν ε, πολλές μελέτες εκεί. Εμείς βασιζόμαστε στην μελέτη McKinsey πέρσι και του ΟΣΑ φέτος, που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα ουσιαστικά, ότι περίπου 15% των θέσεων απασχόλησης θα αντικατασταθεί από την τεχνολογία και ένα της θα επηρεαστεί σημαντικά σε ένα εύρος δεκαετίας από σήμερα. Αυτά είναι τα στοιχεία στα οποία εμείς βασιζόμαστε και δεν είναι τόσο καταστροφικά όσα αυτά που ανέφερε ο προηγούμενος συνάδελφος, αλλά προληπτικά μπορούμε να πούμε ότι αν όλες αυτές οι μελέτες καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτή την υπόθεση. Τρίτον, η μελέτη μας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι, τα, οι φυστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις στο εργατικό και ε, ε, δίκαιο ε, σημειώνουν καθυστέρηση σε σχέση με την πραγματικότητα και το χάσμα αυτό αυξάνεται. Η αγορά εργασίας ε, κάνει τεράστια άλματα και υπάρχει τεράστια ε, διαφοροποίηση και ως προς τις νέες τεχνολογίες, ενώ η νομοθεσία τροποποιείται μόνο οριακά. Αυτό είναι αρνητικό γιατί αυξάνεται το χάσμα και δεν υπάρχει χρόνος. Μας είχε απασχολήσει ιδιαίτερα ο διεθνής αντίκτυπος των όσων ε, ενδεχομένως συμβούν. Και με ενδιαφέρον βλέπουμε ότι το μέλλον της αγοράς εργασίας θα επηρεαστεί από δύο βασικούς παράγοντες. Πρώτον, ε, η τεχνική ηγεσία ε, που έχει σχέση με το επενδυτικό πλαίσιο, δηλαδή ένα νομοθετικό πλαίσιο, θα έλεγα εγώ ως νομικός, που ε, διέπει τον υφιστάμενο επιχειρηματικό ε, κόσμο και δεύτερον η εκπαίδευση που έχει ε, δεσπόζουσα θέση. Στις ΗΠΑ βλέπουμε ότι η Silicon Valley έχει αυτή την ηγετική θέση που βλέπετε σε πράσινο η Ασία εξαρτάται από ορισμένε χώρες για να τα πάει καλύτερα και από την Ευρώπη βλέπουμε από το βορρά προς τον νότο. Δύο είναι οι ήπειροι δυστυχώ που έχουν μείνει πίσω. Η Αφρική και η Λατινική Αμερική που έχουν καθυστερήσει και δεν θεωρούμε ότι θα ε, καταφέρουν να μειώσουν αυτό το χάσμα. Αν δείτε τον παγκόσμιο αντίκτυπο της ψηφιοποίησης, με ενδιαφέρον παρατηρούμε ότι οι χώρες με χαμηλό εργατικό κόστος δεν θα έχουν πλέον αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο μέλλον. Αν δείτε για παράδειγμα την υφαντουργία, ε, το, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κλάδου γίνεται και διεξάγεται στο Βιετνάμ, στο Μπαγκλαντές και στην Κίνα. Όμως βασίζεται στη χειρονακτική εργασία που θα εξαφανιστεί αρκετά σύντομα. Αυτό σημαίνει ότι τα FE, e, λεγόμενα FEE e, ε, εργοστάσια θα επιστρέψουν ε, στις αγορές όπου γίνεται η κατανάλωση, ε, Ευρώπη, Αμερική, ίσως και Κίνα. βασίζονται σε, στα, στο χαμηλό εργατικό κόστος σε μεγαλύτερο βαθμό γι' αυτό. Η μελέτη του 17 της McKinsey τονίζει ότι το ποσοστό των των, των δραστηριοτήτων που θα εκτοπιστούν είναι ε, αυξημένο στις πλούσιες χώρες σε σχέση με τις χώρες μεσαίου και χαμηλού οδήματος. Για παράδειγμα, Ινδία και Κίνα για τα επόμενα δέκα χρόνια τουλάχιστον έχουν χαμηλότερες πιθανότητες ε, να χάσουν πολλές θέσεις εργασίας γιατί αυξάνεται η μεσαία του τάξη. Ε, και έτσι αυξάνεται και η ζήτηση ε, για τον τομέα των κατασκευών και άλλων υπηρεσιών για αυτή τη μεσαία τάξη. Ενώ χώρες όπως οι χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, που γυράσκουν και ως προς το εργατικό του δυναμικό και ως προς τον πληθυσμό τους ευρύτερα, θα χάσουν περισσότερες θέσει εργασία που θα εκτοπιστούν δηλαδή αλλού στο εγγύ μέλλον. Αν δείτε αυτές τις θέσεις εργασίας. Θα υπάρξει μια πόλωση. Θα έχουμε ε, θέσεις εργασίας υψηλής που θα διατηρήσουν τα επίπεδα ανάπτυξή τους, ε, και στις θέσεις εργασίας ε, χαμηλής εξειδίκευσης εκεί υπάρχει μια διχογνωμία. Πράγματι, λιγότερες θέσεις εργασίας θα ε, διατηρηθούν εκεί σε ό,τι φορά τις κατασκευές, όμως για τους άλλους κλάδους όπως είναι τα γυροκομεία, ε, όλος ο κλάδος της παροχής φροντίδας, εκεί θα χρειαζόμαστε περισσότερα χέρια. Αλλά για παράδειγμα, είναι και πολιτιστικό το ζήτημα. Στην Ιαπωνία θα υπάρχουν πολύ περισσότερα ρομπότ που θα φροντίζουν ε, τους ηλικιωμένους. Δεν ξέρουμε πώ ακριβώς θα είναι αυτή η αύξηση, γιατί έχει και πολιτισμικές διαστάσει. Όμως όλες οι μελέτες ε, καταλήγουν ότι ε, στα μεσαία επίπεδα management θα είναι το μεγαλύτερο, ο μεγαλύτερος βαθμός Εκεί μπορεί αυτοί οι εργαζόμενοι όντω να αντικατασταθούν και αρκετά σύντομα από την τεχνολογία, από αλγορίθμους. Έτσι θα έχουμε αυτές τις μεσαίε διοικητικέ θέσει μεσαίου εισοδήματο που θα μπορούν να αντικατασταθούν από την τεχνολογία αρκετά σύντομα και χρειαζόμαστε μία ε, απάντηση για το τι θα απογίνουν όλοι αυτοί. Αν ε, δείτε ποιο είναι το τέλειο σύνολο δεξιοτήτων ε, του εργαζόμενου, του μέλλοντος, βλέπουμε ότι με την εισαγωγή όλων των αλγορίθμων και των ε, ε, λογισμικών και προγραμμάτων ο παλιο παραδοσιακό τρόπος εκμάθησης που όλοι μάθαμε ανήκει στο παρελθόν. Χρειαζόμαστε έναν εργαζόμενο που να επιλύει δύσκολα και περίπλοκα ε, προβλήματα με κριτική σκέψη, με λογική, ε, που μπορεί όμως να εργαστεί και στο πλαίσιο ομάδας, είναι διπλωμάτης, ε, γνωρίζει τις ψηφιακές τεχνολογίες από μικρός και έχει την απαραίτητη ευελιξία για να ε, εργαστεί και να κινηθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο που συνεχώς ε, μεταβάλλεται. Και αυτό ασκεί, θα ασκήσει μεγάλη πίεση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα και στην πρωτοβάθμια και θεωροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στην ίδια την εκπαίδευση των εργαζομένων. Γιατί από τις μελέτες προκύπτουν ότι οι εργαζόμενοι που κατά πάσα πιθανότητα θα αντικατασταθούν στο μέλλον είναι αυτοί που ε, λαμβάνουν ε, λιγότερη επαγγελματική εκπαίδευση άπαξ ε, και μπουν στην αγορά εργασίας. Εάν δείτε τώρα τις δομές των επιχειρήσεων, που είναι αυτό που με απασχολεί εμένα υπάρχουν πολύ ουσιαστικές διαφορές. Έχουμε ε, και νέους όρους ακόμα, όπως το crowd workers. Ε, είναι ένα μεταβαλλόμενο ε, περιβάλλον απασχόλησης. Θα έχουμε ανοιχτή καινοτομία, δομές matrix αντί για ιεραρχία. θα ενισχύονται οι ομάδες έργου αντί να λαμβάνονται απόψεις σε κεντρικό επίπεδο. Το εργατικό μας δίκαιο όμως ε, συνάδει με τον παλαιό κόσμο. Δυσκολεύεται να ακολουθήσει αυτές τις ε, εξελίξεις, γιατί όλοι οι όρκοι και το πλαίσιο που έχουμε ακολουθεί τους παλιούς κανόνες. Έχουμε για παράδειγμα ιεραρχία και κεντρική λήψη αποφάσεων. Εάν να δώσουμε έμφαση τώρα ε, στις ε, ομάδες έργου, τότε υπάρχει και ζήτημα συμμόρφωσης, γιατί με το παλιό σύστημα ένας είναι αυτός που ηγείται του έργου και λαμβάνει και την ευθύνη. Τώρα για το αίσιο τέλος που ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές, όλα αυτά εξαρτώνται από το καλό νομικό σύστημα οι νόμοι δεν πρέπει να είναι αντιδραστικοί. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στον τομέα των υπηρεσιών. Δεύτερον, νομίζω ότι πρέπει να εντοπίσουμε συγκεκριμένους τομείς ε, της νομοθεσίας ε, του 20ου αιώνα, να αλλάξουμε την ε, οδηγία περί ωραρίου, να περιορίσουμε τις 11 ώρες ε, ή και να προβλέψουμε και κάποιες διακοπές, να υπάρχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις, η ρύθμιση de minimis, ε, το άρθρο 23 της ε, μη επαναφοράς, αυτά πρέπει να αναθεωρηθούν. Όσον αφορά τα, την εργατική νομοθεσία, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε εντολή στα κράτη-μέλη να ψηφιοποιήσουν την αντιπροσωπευτική εργασία των εργαζομένων. Αυτό να γίνει υποχρεωτικό, όπως ε, συμβαίνει και στην ε, οδηγία περί κινητικότητας. Η δουλειά των ε, συνδικάτων και των Works Councils των προσώπων των εργαζομένων είναι πολύ περισσότερο ψηφιοποιημένη σήμερα. Εξάλλου, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να υπάρχει και κάποια εκπαίδευση, κυρίως για τους εργαζόμενους με περιορισμένες δεξιότητες και Νομίζω ότι η μελέτη του Πανεπιστημίου του Λίτς στα άτομα στους ε, αυτοαπασχολούμενους για αυτούς προβλέπει κάποια κοινωνικά δικαιώματα, βεβαίω και κάποιες υποχρεώσεις. Καλά όλα αυτά εκτός από τις λογικές συμβάσεις. Εγώ θεωρώ ότι οι ίδιοι θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν αν θέλουν να προσχωρήσουν σε ένα συνδικάτο ή όχι. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι αυτόματα ε, θα πρέπει οι ελεύθεροι επαγγελματίε να καλύπτονται ε, για να ε, καλύπτονται όλοι όσοι βρίσκονται και στην εποχική απασχόληση, εποχική και μερική απασχόληση. Για να ολοκληρώσω, τα έλεγα ότι έχει έρθει η στιγμή για να δραστηριοποιούμε. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να μας ε, κατακυρεύσει αυτό το τσουνάμι που έρχεται. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην επόμενη μιλήτρια, την κυρία Φράνκα Σάλης, η οποία είναι η συγγήτρια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Θα μας μιλήσει για τις νέες μορφές της απασχόλησης, για την πρόοδο και τις δυνατότητες που έχουν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, καλημέρα σας και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρέμβω για τα θέματα αυτά. Καταρχάς, λοιπόν, λαμβάνω τον λόγο εκ μέρους σε ΟΚΕ. Είμαι Γαλλίδα και συμμετέχω στην ε, Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και στο Γαλλικό Συνδικάτο το αντίστοιχο. Η ΕΟΚΕ έχει γνωμοδοτήσει αρκετές φορές για το θέμα της ψηφιοποίησης της εργασίας για τους εργαζομένους, καθώς επίσης και για τις άλλες πλευρές της κοινωνίας των πολιτών, γιατί να υπενθυμίσω ότι εμείς εκπροσωπούμε τους εργαζόμενους εργοδότους, αλλά φυσικά και οργανώσεις καταναλωτών και άλλα μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Καταρχάς να πω ότι η ψηφιοποίηση είναι, ε, και η τεχνητή νοημοσύνη είναι θέματα τα οποία προσφέρουν ευκαιρίες αλλά ενέχουν και κινδύνους. Και επομένως η ΕΟΚΕ δεν είναι αντίθετη σε αυτή την αλλαγή. Δεύτερον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ευρώπη θέλει μια δίκαιη ψηφιακή μετάβαση, η οποία θα βασίζεται στις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τις υπενθυμίσει αυτές τις αξίες, πλήρης απασχόληση, ε, κοινωνική προστασία, υψηλό επίπεδο προστασίας και μείωση της ένδυας και των ανισοτήτων. Και φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχουν τεχνολογικές θέσεις εργασίας πρέπει να είναι χαμηλότερης ποιότητας, να παρέχουν και να δημιουργούν ανισότητες και να μην υπάρχει προστασία. Αυτές λοιπόν είναι οι αρχές οι οποίες ε, ε, διέπουν την όλη ε, ε, διαδικασία. Επίσης, για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί πλήρως την αυτοματοποίηση Ευρώπη και τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά, ανταποκρίνεται στις ε, προκλήσεις για τις δεξιότητες και τα προσόντα, το οποίο αναφέρθηκε αρκετές φορές σήμερα, ένας κοινωνικός διάλογος σε μόνιμη βάση με τους κοινωνικούς εταίρους και κατάλληλες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε και ένα σύστημα ε, φορολόγησης το οποίο να είναι αντίστοιχο των ε, έγιναν αρκετές παρεμβάσεις, ε, επομένως δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία που ακούστηκαν. Οι προβλέψεις ε, συνολικά είναι συγκεκριμένες και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι πιο ευάλωτοι από κάποιους άλλους και θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο ακριβώ αυτέ τι ομάδε ανθρώπων. Και φυσικά όταν αναφερόμαστε στην Ευρώπη, αναφερόμαστε και στα κράτη-μέλη και οι χώρε δεν ε, έχουν ε, κατάλληλη προστασία για του κινδύνου αυτομετοποίηση. Υπάρχουν ε, τελείω διαφορετικά μέτρα και σταθμά. Για παράδειγμα, στη Σλοβακία και στη Φιλανδία ή στην Ορβηγία υπάρχουν διαφορετικές ε, καταστάσεις και πολύ μεγάλες ανισότητες. Και επίσης θα πρέπει να συγκρατήσουμε, και ακούστηκε αυτό, ότι επειδή υπάρχει δυνατότητα αυτοματοποίηση μια θέση εργασία, δεν σημαίνει ότι θα αυτοματοποιηθεί, διότι επισέρχονται και άλλοι παράγοντε και δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Ε, και επομένω ε, υπάρχουν και ε, παράγοντε νομοθεσίε, πολιτικών επιλογών, δημογραφικοί παράγοντε. Για παράδειγμα, αυτοκινητοβιομηχανίε στη Γερμανία υπάρχουν πολύ περισσότερα ρομπέτ, ρομπότ από ότι στην αυτοκινητοβιομηχανία της Γαλλίας. Και γιατί, γιατί ε, στη Γερμανία υπήρχε έλλειψη στη ζήτηση, επομένως υπήρξε αυτοματοποίηση. Αλλά υπάρχουν και θέσεις εργασίας και τομείς οι οποίοι ε, μπορεί να φυγούν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο από την αυτοματοποίηση. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικές διαφορές στα κρατημέλη, διαφορές στα προσόντα και θα πρέπει η Ευρώπη να έχει και κάποιες πολιτικές οι οποίες θα υποστηρίζουν περισσότερο τις χώρες που θα μπορούσαν να πληγούν από την κατάσταση. Σίγουρα υπάρχει η εκπαίδευση και οι δεξιότητες που έχουν σημασία, αλλά σε μια γνωμοδότηση που έχουμε στα σκαριά για την τεχνική νοημοσύνη και την εργασία υπάρχουν τρεις πιθανές λύσεις. Η τεχνητή νοημοσύνη που περιλαμβάνει τους πάντες, να αναφερόμαστε σε κοινωνικές και υπεύθυνε αναδιαρθρώσεις, γιατί είναι αναπόφευκτο να γίνει αναδιάρθρωση. Και τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη που να περιλαμβάνει τους πάντες. Αυτό σημαίνει ότι ε, βάσει του μοντέλου, για παράδειγμα, των κάτω χωρών, θα πρέπει να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι, γιατί ο κόσμος της εργασίας είναι πολύ σημαντικός ε, για όλες αυτές τις αλλαγές και επομένως θα πρέπει να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην εισαγωγή αυτών των αλλαγών να τους εμπλέξουμε, να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δεξιότητές τους ε, σε συνδυασμό με έξυπνα μηχανήματα και φυσικά θα πρέπει να μένουν και στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας και να συμμετέχουν και στη βελτίωση. Ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η αρχή. Μία τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν που θα περιλαμβάνει τους πάντες χωρίς αποκλεισμούς και να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Επίσης υπάρχουν οι αρχές της διαφάνειας ε, και των ευθυνών που η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πρόσφατα συμπεριέλαβε στη δέσμη μέτρων για τη τεχνητή νοημοσύνη και νομίζω ότι αυτή η αρχή της διαφάνειας, της ισότητας και της υποφθηνότητα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και στον κόσμο και να έχουμε φυσικά δίκαιες αρχές. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει ε, να... Ε, ε, στερούμε από τους εργαζομένους την εργασία τους. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να σκεφτούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα υπόκειται σε ένα μηχάνημα. Και επίση ε, να προβλέψουμε. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Διότι αν κάνουμε πράγματα καθυστερημένα και ήδη έχουμε καθυστερήσει, ε, τότε θα υποστούμε απλώ τι συνέπειε και δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι τόσο γρήγορε αλλαγέ. Όσον αφορά την υπεύθυνη διαχείριση των, της Αναδιαμόρφωση σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μην χάσουν τις εργασίες τους, να γίνεται η μετάβαση, η αλλαγή και επίση υπάρχει και καινοτόμος ε, κοινωνική προσαρμογή. Γίνεται ένας κοινωνικός διάλογος, ο οποίος αρχίζει για παράδειγμα και ανατομή. Στη Γαλλία υπήρχε το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Δηλαδή, ότι τα τεχνολογικά μέσα που έχουν στη διάθεση οι εργαζόμενοι, επειδή μπορεί να παρέχονται ανα πάσα στιγμή και να υπάρχει υποχρέωση να είναι κάποιο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο ανα πάσα στιγμή, να απαντά σε email, ε, στο τηλέφωνο, σε οτιδήποτε. Υπάρχει ένα νέο νόμο λοιπόν, ο οποίο αρχίζει σιγά σιγά να έχει κάποιο αντίπτυκο όπω στην Ευρώπη. Επίση, πρέπει να ε, δίνουμε ε, σημασία την ατομικότητα, στο πρόσωπο, διότι ε, μπορεί κάποιος να έχει διαφορετικές ιδιότητες, να είναι εργαζόμενος, αυτοαπασχολούμενος κλπ. Κάθε φορά που αλύζει ε, θα πρέπει να ε, τον συνοδεύουν και τα δικαιώματά του, δικαίωμα στην προστασία, κοινωνικά επιδόματα κλπ. Και τέλος, Υπάρχει και το θέμα, για παράδειγμα, το οποίο προέκυψε πρόσφατα στη Δανία. Υπήρχε ε, συλλογική διαπραγμάτευση για συμβάσει εργασία με μια πλατφόρμα τεχνολογική. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει προσαρμογή, είναι στο δημόσιο τομέα τη ιδιοκτησία και υπάρχει μια συμφωνία διάρκεια ενό έτου και μετά θα επανεξεταστεί, αλλά λαμβάνει υπόψη τι νέε μορφέ εργασία και επειδή κάποιο εργάζεται σε μια πλατφόρμα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να του στερούμε τα δικαιώματά του. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να προσέξουμε και τα όσα συμβαίνουν. Τα συνδικάτα βεβαίως ε, θα πρέπει να καινοτομήσουν. Ε, δεν προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα με την ε, ταχύτητα της τεχνολογίας η οποία σίγουρα κάνει ελματώδη Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και κάποια πράγματα και αυτό είναι σημαντικό και θεωρώ ότι η τεχνική τη νοημοσύνη θα βοηθήσει και τα συνδικάτα για τα μέλη και για τους εργαζομένους μισθωτούς ή μη. Θα σταματήσω εδώ βεβαίως και ευπρόσδεκτες τυχόν ερωτήσεις από πλευρά σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εάν λοιπόν θέλει κάποιος ε, να υποβάλει κάποια ερώτηση στους ε, ομιλητές, ε, παρακαλώ, βεβαίως έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε ερωτήσεις. και πραγματικά πρέπει να πω ότι είναι λιγάκι απογοητευτικό το όλο αυτό που μας παρουσιάσατε. Εγώ σημείωσα κάποια πράγματα. Είπατε ότι θα είναι δύσκολο για τους ενδιαφερόμενους να βρουν θέση απασχόλησης, να διατηρήσουν αυτή τη θέση, γιατί θα πρέπει συνεχώς να αποκτά κανείς ε, νέες δεξιότητες, ε, νέα προσόντα. Ε, η τεχνική επανάσταση πράγματι ασκεί αρκετά μεγάλη πίεση στο χώρο εργασίας ή όπου, εν πάση περιπτώσει, βρίσκεται κανείς. Ακούσαμε επίσης ότι η νομοθεσία δεν είναι επικαιροποιημένη όσον αφορά αυτή τη νέα αγορά εργασίας και τις νέες τεχνικές. Ακούσαμε ότι θα διευρύνεται όλο και περισσότερο το χάσμα ανάμεσα σε διάφορους ανθρώπους ε, ανάλογα αν έχει κανείς ε, καλή εκπαίδευση, αν έχει μέτρια, αν ε, δεν έχει καθόλου εκπαίδευση. Σας είπα το ε, χάσμα θα γίνεται όλο και μεγαλύτερο και θα προκύπτουν όλο και πιο ε, σκληρές συγκρούσεις. Πρέπει κανείς ε, να είναι ευέλικτος καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, στον χώρο εργασίας. Πρέπει να είναι ελκυστικός στην αγορά εργασίας και αν είναι κανείς αυτοαπασχολούμενος θα πρέπει να αρέσει τουλάχιστον στον εαυτό του για να μπορεί να είναι να παραμένει προσιλωμένος ε, στο στόχο του. Βεβαίω ε, δεν μπήκατε σε λεπτομέρειε ε, για το τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει τεχνική επανάσταση στο χώρο της φορολογίας. Όμως η εικόνα είναι ζωφερή θα έλεγα. Τα συζητάμε βέβαια αυτά κατά καιρού στην Επιτροπή μας αλλά και σε άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι πάντα έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή όταν προκύπτει μία μεγάλη αλλαγή φοβόμαστε την αλλαγή αυτή και παράλληλα υπάρχει και η νέα γενιά η οποία βέβαια ε, αγκαλιάζει κάποια στοιχεία αυτής της αλλαγής. Σε τελική ανάλυση τι πρέπει να κάνουμε. Ε, δεν ξέρω πώς πρέπει να προχωρήσουμε ως ε, ερευνητές, ε, ως συνδικάτα, ως εργατικά συνδικάτα, ως ε, βουλευτές. Δεν ξέρω ε, πώς μπορούμε να βρούμε ένα τρόπο έτσι ώστε οι άνθρωποι να νιώθουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητες που έχουν, στις δυνατότητες να εντάσσονται στο χώρο εργασίας και να εντάσσονται υπερήφανοι στον, στο εργατικό δυναμικό. Και αυτό να ισχύει και για, μετά από 10-15 χρόνια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Και εγώ σκεφτόμουν, να ξέρετε, σκεφτόμουν τελικά αυτά που άκουσα ήταν ε, θετικά ή αρνητικά. Αυτό λέει βέβαια κάτι και για μένα, ε, το πώς πρέπει να χωρίζω τα πράγματα. Γιατί ε, σε τελική ανάλυση θεωρώ ότι πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα, ένα μείγμα μηνυμάτων. Ε, οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης έχουν προβλεφθεί εδώ και αρκετό. Έχουμε τώρα τις μελέτες της McKinsey και του ΩΣΑ που ίσως να μην προβλέπουν την πλήρη ε, πόλωση της αγορά εργασίας. Σας λέω, υπάρχει ένα αμάλγαμα μηνυμάτων. Και διερωτήθηκα ε, μήπως ισχύει εδώ ε, αυτό που ισχύει με την κότα και το αυγό. Κατά κάποιον τρόπο όλες αυτές οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις ε, δεν μπορεί κανείς ε, να είναι πάντα στο χώρο εργασίας, ε, μπορεί να κάνει τη δουλειά του αρκετά ανεξάρτητα και τελικά αυτό να είναι και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα από το να είναι κανείς στο χώρο εργασίας και να έχει συνέχεια πάνω από το κεφάλι του τον εργοδότη. Ίσως λοιπόν ε, να χρειαζόμαστε και λιγότερους ε, μεσαίους, ε, μεσαία διευθυντικά στελέχη, τα οποία να εποπτεύουν διαρκώς ε, την εργασία. Αυτό όμως που με ανησυχεί εμένα πάνω απ' όλα είναι το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση πράγματι καθιστά σαφές ότι το χάσμα ανάμεσα στην πραγματικότητα και, το χώρο, και, τον, και την εργατική νομοθεσία ε, ότι ανάμεσα δύο υπάρχει μια μεγάλη διαφορά και εσείς μιλήσετε για ένα επερχόμενο τσουνάμι και κατά κάποιον τρόπο υπάρχει και ένα μεγάλο οικονομικό πλεονέκτημα στο να χρησιμοποιεί κανείς την ε, ψηφιοποίηση Χρησιμοποιώντας ε, την ε, ψηφιοποίηση κατά κάποιον τρόπο υφαρπάζουμε την προστασία από τους εργαζόμενους. Γιατί αν ο εργαζόμενος, παραδείγματος χάρη στην Uber, δεν είναι πια απασχολούμενος με εξαρτώμενη σχέση απασχόληση, αλλά αυτό απασχολούμενος, ε, καλείται και ο εργαζόμενος αυτός να καταβάλει τις εισφορές του στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Εγώ θέλω να ρωτήσω, οι όταν περνάνε από μισθωτή, από το μοντέλο του μισθωτού στο μοντέλο του από αποσχολούμενου, αυτό είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο. Σήμερα ε, και στην έκθεσή σας ε, αναφέρεται παραδείγματο χάρη ότι υπάρχουν εταιρείε όπω η McDonald's που δεν καταβάλουν του προβλεπόμενου μισθού στου εργαζόμενου και δεν καταβάλουν και τι τις ε, ε, προβλεπόμενε εισφορέ. Φοροδιαφεύγουν. Κατά κάποιον τρόπο λοιπόν πώ μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το τσουνάμι ή πώς ε, μπορούμε να αποφύγουμε την καθυστέρηση στην εργατική νομοθεσία. Η ευρωπαϊκή πρόταση για αυτό που αποκαλείται, δεν θυμάμαι καλά να σας πω λέει ομιλήτρια, Κάπως ε, μου ξεφεύγει τώρα, δεν, δεν τα θυμάμαι και αυτό δεν είναι προσωπικό μου πρόβλημα, το πρόβλημα των διαφανών και προβλεπόμενων συνθήκων εργασίας. Το βρήκα. Λοιπόν, αρκεί αυτό για να αποφύγουμε το τσουνάμι και οι εταιρείε οι οποίες έχουν πολλά οικονομικά ωφέλη χρησιμοποιώντας την ε, τεχνολογία για να αφαιρέσουν από τους εργαζόμενους τα εργατικά τους δικαιώματα, πώς μπορούμε να τις ε, καλέσουμε στην ε, τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει σε επίπεδο κράτους μέλους ή πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλιστα, πολλά ερωτήματα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, δείξατε πολλά ζητήματα. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Δεν νομίζω ότι η πρόταση που βρίσκεται τόσο θα επιλύσει το ζήτημα της οικονομίας πλατφόρμας. Ίσως να λύσει το ζήτημα των επισφαλών σχέσεων εργασίας, όπου θεωρούμε ότι δεν έχουν εκχωρηθεί τα ε, απαραίτητα δικαιώματα στους εργαζομένους. Περισσότερο λοιπόν στρέφεται προς το παρελθόν παρά προς το μέλλον. Από την μελέτη του Πανεπιστημίου του Λίτς προκύπτει ότι ακόμα και η προστασία σε ό,τι αφορά... Πρέπει να, να δώσουμε σε αυτούς τους εργαζόμενους ε, δικαιώματα υπό την κοινωνική προστασία και μάλιστα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να έχουν λοιπόν τη δυνατότητα το ένα δικαίωμα να πάει προς το επόμενο. Γιατί ο κάθε εργαζόμενος θα εργάζεται για διαφορετικές οντότητες, διαφορετικούς φορείς. Και αν δείτε τα επιμέρους ε, μοντέλα απασχόλησης ε, Ισπανία, Ηνωμένου Βασιλείου, κάποιοι λένε ότι επιπλέον των ε, δικαιωμάτων κοινωνικής προστασίας υπάρχουν και κάποια δικαιώματα υπαλλήλων, όπως είναι οι διακοπές ή ο βασικός μισθός, που θα πρέπει να δοθεί και σε αυτούς. Νομίζω ότι αυτό είναι ο σωστός τρόπος, γιατί έτσι έχουμε ίσους όρους για όλους και είπατε ότι μπορεί να το εξοποιήσουν ε, γενικά να αξιοποιήσουν αυτή τη νέα δυνατότητα οι εταιρείε ε, για να ε, φοροδιαφύγουν. Έτσι λοιπόν κάπως αμπλύνεται αυτός ο κίνδυνος, αυτό το πρόβλημα. Συχνά ακούμε για τη λεγόμενη χαμένη γενιά. Για παράδειγμα, ο διανομέας ή ο ταμείας ε, του σούπερ μάρκετ. Έχουμε εκατομμύρια εργαζόμενους στον τομέα του λιανικού εμπορίου και ε, της υλικοτεχνικής υποδομής και ξέρουμε ότι ήδη υπάρχουν αυτές οι τεχνολογίες που θα φέρουν τα πάνω κάτω. Επομένω, πρόκειται για εκατομμύρια θέσει εργασία που μπορούν να χαθούν και δεν νομίζω ότι ο ε, σημερινός διανομέας θα γίνει προγραμματιστής αύριο. Πρέπει λοιπόν εκ των προτέρων να υπάρξει πολιτική παρέμβαση. Γιατί υπάρχουν ε, αφενός και επισφαλείς θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή και μπορούμε αυτό να διορθώσουμε. Από την άλλη υπάρχουν κλάδοι ε, και θέσεις εργασίας που ξέρουμε ότι θα χαθούν. Για μας ε, είναι σχεδόν δεδομένο αυτό. Ευχαριστώ κύριο Σέγγλωμ, έχει Ευχαριστώ πολύ. Πρώτον, κατά πόσο πρόκειται για ε, θετικό ή αρνητικό αφήγημα. Όπως και να έχει είναι ένα αφήγημα. Αν δείτε τις ε, ε, εκτιμήσεις του ΟΣΑ, αναφέρεται ένα ποσοστό του 15% που θα χαθούν και άλλο 10-15% που θα αλλάξουν μορφή. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με στοιχεία που δεν διαφέρουν σε σχέση με αυτά που έχουμε δει και εμείς ε, στη ζωή μα. Και ο 20 ο αιώνα, για παράδειγμα, στην Ευρώπη επέφερε τεράστιε αλλαγέ και στην αγορά εργασία. Τεράστιε ε, δομικέ αλλαγέ και ερχόμαστε αντιμέτωποι με αυτό. Με τι κατάλληλε πολιτικέ μπορούμε να το κάνουμε και αυτό είναι και το θέμα τη συζήτηση. Πώ θα γίνει αυτό. Βέβαια, το ερώτημα δεν είναι πώς θα επιβραδύνουμε αυτή την μεταβολή, αλλά πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι θα καταφέρουν να, τα, να αντεπεξέλθουν σε, αυτή τη, σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο. Ε, γίνεται αυτό με τη διαβίου μάθηση και κατάρτιση, αλλά θα πρέπει και να ε, υλοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες με έναν τρόπο που να αισθάνεται και ο κόσμος ότι έχει λόγο. Και πάλι επανερχόμαστε στο ζήτημα της ε, ε, διαβούλευσης, το οποίο μπορεί να γίνει πλεονέκτημα για την Ευρώπη. Τώρα, κατά πόσο η εργατική νομοθεσία έχει μείνει πίσω. Είναι επικίνδυνη αυτή η έννοια. Γιατί και πάλι ο 20 ο αιώνας μας έχει διδάξει ότι η εργατική νομοθεσία ήταν ιδιαίτερα ευέλικτη και βασικές αρχές του εργατικού δικαίου, όπως η έννοια του υπαλλήλου, έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εξελίσσονται όταν εξελίσσεται και η κοινωνία και η οικονομία. Αν αρχίσουμε να λέμε συνεχώς ότι η εργατική νομοθεσία έχει μείνει πίσω, ξανά και ξανά, τότε αυτό θα αρχίσει να ισχύει. Από την άλλη πρέπει να προσπαθούμε ε, κάπως να καθιστούμε πιο ευέλικτες τις έννοιες που έχουμε. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες ακόμα εξαρτώνται ε, στο από το αφήγημα που πουλάνε προς τους επενδυτές και πρέπει εμείς πάντα με κριτική ματιά να εξετάζουμε αυτή την επιχειρηματολογία. Και τώρα, στο επιχειρηματικό μοντέλο της εξαίρεσης ε, εργαζομένων από συγκεκριμένα δικαιώματα, εδώ και πάλι βλέπουμε τους ε, οδηγούς, για παράδειγμα, που ε, ταξινομούνται είτε ε, υπό το καθεστώς των υπαλλήλων, είτε προς τον αυτοπασχολουμένων. Η φορολογία εδώ είναι πολύ σημαντικός φορέας. Έχουμε δει ότι ε, ξαφνικά μπορεί κάποιος να προσλάβει κάποιον για λιγότερα χρήματα. Το σημαντικό λοιπόν είναι εδώ η φορολογία και ε, οι εργοδοτικές εσφορές για αυτούς τους υπαλλήλους να είναι πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε και πάνω κάτω τα ίδια δικαιώματα για τους υπαλλήλου και τους αυτοαπασχολούμενους. Πρέπει να αρχίσουμε να εξετάζουμε τις σταδιοδρομίες αυτών των εργαζομένων. Πρόκειται δηλαδή για ένα εφαλτήριο για αυτούς τους εργαζομένους ή περιστασιακή αυτή απασχόληση ή απλώς ξεμένουν εκεί. Συνήθως δυστυχώς βλέπουμε ότι όσο πιο επισφαλής είναι η θέση εργασίας από την οποία ξεκινάει αυτός ο υπάλληλο, ο εργαζόμενος, τόσο πιο ε, δύσκολα θα τα βρει και στην πορεία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο καθηγητής Βαλέριο Δεστέφανο, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να περιμένετε να βλέπετε καθαρά αρνητικέ ή καθαρά θετικέ συνέπειε ε, της τεχνολογική εξέλιξη των χώρο εργασία. Διότι όλα αυτά προκύπτουν από ε, το γεγονός ότι θεωρούμε ότι είναι κάτι εξαιρετικό η τεχνολογία και ότι συμβαίνουν μόνο καλά ή μόνο άσχημα πράγματα. Στην πραγματικότητα η τεχνολογία είναι τμήμα της ζωής, υπάρχουν και καλά και κακά και η νομοθεσία υπάρχει για να προσπαθήσει να ρυθμίσει τα πράγματα και να εξασφαλίσει ότι η πραγματικότητα θα πάει σε καλύτερη κατεύθυνση από αυτή που θα είχαμε χωρίς νομοθεσία. Τώρα, όσον αφορά το ερώτημα για το πώς θα πείσουμε τις πλατφόρμες να καθίσουν γύρω από ένα τραπέζι και ούτω καθεξής. Σε πολλές περιπτώσεις το πρόβλημα είναι ότι δεν χρειάζεται να τους πείσουμε. Κάθε επιχείρηση, κάθε ε, ε, οργανισμός πρέπει να συμμορφωθεί με συγκεκριμένους κανόνες. Και όταν δεν είναι συμβατά με την κείμενη νομοθεσία, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι και τα επιχειρηματικά μοντέλα ε, φτιάχνονται για να παρακάμψουν τον νόμο και επομένω αυτό δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται. Δεν ισχύει βέβαια πάντα αυτό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείε ε, πραγματικά ε, χρησιμοποιούν το γεγονός ότι δημιουργούν διαταραχές, αλλά στην πραγματικότητα η μόνη διαταραχή που προκύπτει είναι ότι ε, απασχολούν κόσμο χωρίς να αναλαμβάνουν και το τίμημα η τεχνολογία, ε, επίσης λέμε ότι θα χρησιμοποιείται μόνο για να γινόμαστε περισσότεροι αυτόνομοι. Δεν ισχύει αυτό. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγχουμε και τις επιδόσεις στην εργασία πιο στενά. Και αυτό γίνεται όχι μόνο στην οικονομία πλατφόρμας, αλλά και στις πιο παραδοσιακές μορφές ε, ε, οικονομίας. Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν βραχιολάκια για να παρακολουθείτε πώς ε, ε, εργάζεται κάποιος ή για να δει τη διάθεσή του ανάλογα με τις ε, διακυμάνσεις στη φωνή και ούτω καθεξής. Και όλα αυτά σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι θετικό διότι μπορεί να βοηθήσει και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία αλλά μπορεί να υπάρχει και εκμετάλλευση των προσωπικών μας δεδομένων και επομένω να είναι αρνητικό σε αυτή την ε, περίπτωση. Δεν υπάρχει δηλαδή άσπρο μαύρο. Θα πρέπει η νομοθεσία να ε, ρυθμίσει τα φαινόμενα αυτά για να αποφύγουμε καταχρήσει. αλλά ταυτόχρονα να υποφεληθούμε και των ευκαιριών που προσφέρει η τεχνολογία. Και αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρολάνο, συνάδελφος. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο πτυχές, οι οποίες θα ήθελα να θίξω εγώ, που νομίζω ότι ε, δεν αναφέρθηκαν επαρκώς ή δεν αναφέρθηκαν κατα, καταλήλως η ψηφιοποίηση παρουσιάστηκε ως κάτι το φυσιολογικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχουν εποχές, υπάρχει άνοιξη, επομένως υπάρχει και τεχνολογική εξέλιξη και ε, πρέπει λοιπόν να διαχειριστούμε μόνο τις συνέπειες. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των ε, τεχνολογικών επιλογών που γίνεται και το θέμα των τεχνολογικών επιλογών θεωρώ ότι είναι θεμελιωδώς πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή αφορά ε, τον τρόπο της κοινωνίας στην οποία θέλουμε να ε, ε, κινούμαστε. Θέλουμε να ε, είμαστε μοχλοί αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Προτείνουμε για παράδειγμα να υπάρχουν ε, ε, μπάτζ σήματα μαγνητικά ε, για να υπάρχει περισσότερο ή κάποιοι οι οποίοι φορούν συνεχώς ακουστικά και αντιδρούν απλώς σε έναν αλγόριθμο και αυτό φυσικά δεν είναι μόνο οι τεχνολογίες καθημερινότητας. Βλέπουμε για παράδειγμα στις αυτοκινητοβιομηχανίες με πιο απλές τεχνολογίες Ε, και ουσιαστικά ο άνθρωπος εκεί έχει γίνει ένα τμήμα της μηχανής ε, στη διαδικασία αυτοματοποίησης. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο θα πρέπει να το δει η κοινωνία όσον αφορά τις επιλογές που κάνουμε στην τεχνολογία και όχι πώς προσαρμοζόμαστε στις επιλογές που έχουν κάνει άλλοι. Δεύτερον, υπάρχει το θέμα του κίνδυνου και της ευκαιρίας ε, Σίγουρα βέβαια θα πρέπει να ε, περιορίσουμε τους κινδύνους και να σταθούμε στις ευκαιρίες, αυτό είναι δεδομένο, αλλά υπάρχει και το θέμα της θέσης του ατόμου, δηλαδή του εργαζομένου στην όλη διαδικασία. Αναφέρθηκατε στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ και το θέμα της ε, ε, του γεγονότος ότι ο εργαζόμενος δεν κατέχει πλέον την εργασία του. Ε, και υπάρχουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες ήδη ε, ε, τις βλέπουμε σήμερα και υπάρχει εξατομίκευση της εργασίας τη διαδικασία της εργασίας και υπάρχουν και συνέπειες φυσικά για την υγεία. Βλέπουμε για παράδειγμα κάποια πράγματα σε θέματα υγείας και ασφάλειας στον τομέα της ε, ε, της εργασίας, ε, υπερκόπωση, αλλά όχι μόνο υπερκόπωση, αλλά και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχουν και νέες ασθένειες επαγγελματικές και φυσικά αυτό σημαίνει ότι χάνεται η αίσθηση της εργασίας για τον εργαζόμενο και ταυτόχρονα υπάρχει και ένας αποκλεισμό από το συλλογικό της εργασίας. Δεν ξέρω λοιπόν αν στη μελέτη σας ασχοληθήκατε με τα θέματα αυτά. Παρακαλώ. Μπορώ να απαντήσω. Η κυρία Σαλής Μαντίνιε. Έχετε δίκιο. Η πρόκληση για τις κοινωνίες μας, η πρόκληση για τις πολιτικές μας και η πρόκληση και των κοινωνικών εταίρων είναι να επιλέξουμε σε ποιο κόσμο θέλουμε να ζήσουμε και τι ρόλο θέλουμε να προσδώσουμε στην ε, τεχνητή νοημοσύνη, στο έξυπνο μηχάνημα και αυτό σήμερα νομίζω ότι δεν έχει απαντηθώ, δεν, δεν έγιναν αρκετές διαβουλεύσεις ε, και δεν έχουν γίνει αρκετές συζητήσει επ' αυτού. Εγώ πιστεύω ότι από πλευράς κοινωνικών εταίρων η διαπραγμάτευση δεν είναι σε αρκετά ικανοποιημένο επίπεδο στην Ευρώπη. Υπάρχει κοινωνικός διάλογος, αλλά τι αποτελέσματα έχει. Μπορώ να μιλήσω λίγο πιο άμεσα και ειλικρινά εδώ. Και νομίζω ότι υπάρχουν αντιστάσεις ε, στη διάθεση να νομοθετήσει και να ρυθμίσει κανείς. Να σας δώσω ένα τελευταίο πρόσφατο παράδειγμα. Η οδηγία γιατί ε, συνθήκες ε, πρόβλεψης της διαφάνειας ε, στην εργασία υπάρχει υποχρέωση να υπάρχει οδηγία γιατί η συλλογική διαπραγμάτευση απέτυχε. Υπάρχει λοιπόν όλος προβληματισμός και πιστεύω ότι στην Ευρώπη δεν είμαστε στο ύψος αυτών που έχει σχεδιάσει η Ευρώπη στην ιστορία της σε επίπεδο αυτονομίας και συλλογικής διαπραγμάτευσης για να ρυθμίσει όλες τις μορφές εργασίας και καινοτομίας σίγουρα είναι πιο εντυπωσιακά όσα βλέπουμε, διότι ε, φανταζόμαστε ανθρωπόμορφα ρομπότ που αντικαθιστούν ανθρώπους κλπ. Αλλά ε, ο όλος προβληματισμός της εισαγωγής της νέας τεχνολογίας και τι συνέπειες έχει για την εργασία, για την ποιότητα, για την οργάνωση της εργασίας και τις συνθήκες εργασίας, της ασφάλειας και της υγείας, είπατε πολύ σωστά κύριε Ρολά, δεν λαμβάνεται δεόντως υπόψη ε, καθολικά ε, αλλά ε, και ατομικά, διότι οι επιχειρήσεις και οι διάφοροι κλάδοι φυσικά έχουν τις διαφορές τους, δεν είναι όλα ίδια και ε, υπάρχει όμως και ένα σοκ το οποίο είναι καθολικό. Ε, το σοκ του απόλυτα καινούριο, όπως το αποκαλούμε στην ΕΟΚΕ. Υπάρχουν, θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ευρωπαϊκό δίκαιο και θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές τις αλλαγές. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτές οι αλλαγές, οι επιλογές, συγγνώμη, λείπουν ε, και υπάρχει και μια πρόσφατη μελέτη του κ. Βιλάνη στη Γαλλία, ο οποίος θέλει να δώσει μια, μια ένα νόημα στην ε, τεχνητή νοημοσύνη και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να προσανατολίσουμε προς αυτό που θέλουμε να γίνουμε αύριο. Και κεντρικό ρόλο φυσικά θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος και η σχέση του με το μηχάνημα. Και ε, σε μια γνωμοδότηση που είχαμε πέρσι για την τεχνητή νοημοσύνη, λέμε ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει τα ενία. Ο άνθρωπος θα πρέπει να μπορεί να ε, χειρίζεται το μηχάνημα. Και αυτό φυσικά το οποίο φοβίζει είναι τα περιβόητα μαύρα κουτιά, δηλαδή αλγόριθμοι οι οποίοι δημιουργούνται και παράγονται χωρίς να γνωρίζουμε ακριβώς τα αποτελέσματά τους. Και νομίζω ότι θα πρέπει να καταρτήσουμε τους, μηχανισμούς μας, ε, τους μηχανικούς μας για τις ε, δεοντολογικές προκλήσεις και τα μηχανήματα τα οποία θα δημιουργήσουμε να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και της ανθρωπότητας. Μπορούν να προσφέρουν μεγάλο καλό σε πάρα πολλούς ανθρώπους, ανθρώπους για παράδειγμα που μπορεί να έχουν μια αναπηρία, ε, κινητική αναπηρία, αλλά φυσικά και όλες τις ευκαιρίες που μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, σε διαγνωστικό επίπεδο, σε επίπεδο υγείας, ε, στην ιατρική. Υπάρχουν ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει να τις ελέγχουμε εμείς. Και όπως πολύ σωστά είπατε, πολύ σωστά κύριε Ρολά, θα πρέπει να υπάρχουν οι μέγιστες δυνατές ευκαιρίες και οι κίνδυνοι, οι αρνητικές συνέπειες να αντιμετωπιστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Να προετοιμάσουμε δηλαδή για αυτό το σενάριο και αυτό σημαίνει να προετοιμάσουμε τον κόσμο του αύριο στον οποίο επιθυμούμε να ζήσουμε. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ, ο Σαντεστέφανο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω στον ε, πιθανό ρόλο της νομοθεσίας, γιατί αναφέρθηκε προηγουμένως ότι κατά καιρού θεωρούμε ότι αυτό θα συμβεί ανεξάρτητα το τι θέλουμε εμείς, δεν έχουμε καμία δυνατότητα παρέμβασης και αυτό είναι δεδομένο το βλέπουμε και στην ίδια ρητορική για την ε, αυτοματοποίηση, για τις θέσεις εργασίες που θα χαθούν, οι νέες τεχνολογίες που θα εισαχθούν ε, θα εκδιώξουν εργαζομένους από την αγορά εργασίας, αλλά ξεχνούμε ως Ευρωπαίοι ότι έχουμε κάποια μέσα ε, στη διάθεσή μας για την διαχείριση των μαζικών απολύσεων και της μαζικής ανεργίας. Έχουμε οδηγία για τις συλλογικές μαζικές απολύσεις που διέπει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ε, εργοδοσίας και εκπροσώπων των εργαζομένων όταν έχουμε να κάνουμε με την αυτοματοποίηση, ε, την απόλυτη συνεργασία κτλ. Αυτό συχνά το ξεχνάμε. Ποτέ δεν ε, λέει κανείς ότι ουσιαστικά ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να αξιοποιηθεί για να έχουμε καλύτερη διαχείριση της αυτοματοποίησης. Και νομίζω ότι ο κοινωνικός διάλογος επίσης θα μπορέσει να συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας και για τι ε, θέσει που θα χαθούν λόγω τη αυτοματοποίηση, αλλά και για τι υπόλοιπε που δεν θα χαθούν. Πώς θα τις ε, χειριστούμε, πώς θα διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία αξιοποιείται προς όφελος ε, όλων και όχι για την πιο στενή επίβλεψη και παρακολούθηση των εργαζομένων. Γιατί και πάλι, αν δεν το κάνουμε αυτό, ε, ο κόσμος θα αρχίσει να φοβάται την τεχνολογία, θα ε, αντιδρά αρνητικά σε αυτές τις αλλαγές και αυτό θα επηρεάσει αρνητικά και την παραγωγικότητα και το ε, οικονομικό όφελος. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κέρια σημασίας να δούμε τα ωφέλη του ευνομοθετήν ως προς την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Έγκμπλουμ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ κέριο αυτό το ερώτημα, κατά πώς πρέπει να αποδεχθούμε την τεχνολογία. Όχι. Εμείς ως άνθρωποι ε, καταδυναστεύουμε αυτές τις τεχνολογίες. Από την άλλη, σε μια ήπειρο όπως η Ευρώπη, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η τεχνολογία είναι ένα από τα πράγματα που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να είμαστε κατά το δυνατόν πιο ανταγωνιστικοί και να δημιουργήσουμε τον πλούτο που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε τη ζωή που θέλουμε. Είναι λοιπόν ένα πολύ καλό επιχείρημα για να είμαστε θετικοί ως προς την τεχνολογία. Από την άλλη πρέπει να δούμε πώς ε, ρυθμίζεται ε, αυτή η τεχνολογία. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση της τεχνολογίας, αλλά των αποτελεσμάτων της. Για παράδειγμα, ε, τεχνητή νοημοσύνη στις διαδικασίες πρόσληψης. Η διάκριση, ε, οι διακρίσει στον τομέα των προσλήψεων δεν επιτρέπονται βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου. Και βέβαια, αν ένα εργοδότη ε, αξιοποιήσει ένα εργαλείο το οποίο προβαίνει στι διακρίσει, αυτό απαγορεύεται. Αν δείτε τώρα ε, την υγεία και ασφάλεια εργαζομένων, συμφωνώ ότι υπάρχουν ανησυχίες εάν κάποιος στο εργασιακό του περιβάλλον δεν έρχεται σε επαφή με τον εργοδότη του, αλλά με ένα ψηφιακό μέσο. Αυτό σαφώς και δημιουργεί διαφορετική εργασιακή σχέση και αυτό αποτελεί κίνδυνο στην εργασιακή σχέση, γιατί ξέρουμε πόσο σημαντική θέση έχουν ε, τα ηγετικά στελέχη, οι μάνατζερ σε σχέση με τον υπάλληλο. Δεν θα πρέπει να χαθεί λοιπόν αυτό και δεν θα πρέπει να βλέπουμε την τεχνολογία ως ε, κάτι το μυθολογικό σχεδόν. Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος πίσω από την τεχνολογία, υπάρχει ένας εργοδότης που ε, χρησιμοποιεί την τεχνολογία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να χαθεί και το θέμα της ευθύνης. Και δεν θα πρέπει να είναι σε θέση ο εργοδότης να κρύβεται πίσω από την τεχνολογία. για να ε, ισχυριστεί ότι ο ίδιος δεν φέρει ευθύνη έναντι των εργαζομένων του. Επομένως, στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουμε μια θετική στάση ως προς την τεχνολογική αλλαγή, γιατί, όπως είπα, αυτό θα δημιουργήσει τον πλούτο που χρειαζόμαστε για το μέλλον μας. Όμως, παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα ε, μοναδικά ενδεχομένω μέσα που έχουμε σε αυτή την Ήπειρο για να ρυθμίσουμε αυτές τις τεχνολογίες. Και πολύ σωστά τα ανέπτυξε αυτά ο Βαλέριο. Ευχαριστώ κύριο Ντάξ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τους συναδέλφους εδώ. Σαφώς και η τεχνολογία δεν είναι θεόσταλτη, ε, αποτελεί αντικείμενο της ανθρώπινης ε, δράσης και διάδρασης. Δημιουργείται λοιπόν, δεν προκύπτει εκ του μηδενός. Όμως ε, να σταθώ σε κάτι άλλο ε, που θεωρώ αρνητικό σε αυτή την ευρύτερη συζήτηση. Εδώ υπάρχει ένα ε, κενό. Αφενός, μπορούμε να πούμε πολλά για τις πιθανές απώλειες. Ξέρουμε τα επαγγέλματα που κινδυνεύουν ε, να αντικατασταθούν από την τεχνολογία. Έχουμε λοιπόν μια καλή εικόνα των επαγγελμάτων και των θέσεων εργασίας που μπορεί να χαθούν. Και αυτό εμπεριέχεται και σε όλες τις μελέτες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Όμως, αυτές οι μελέτες δεν μας λένε απολύτως τίποτα για τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως να δημιουργηθούν από τις νέες τεχνολογίες. Δεν μας λένε τίποτα για τα πιθανά ωφέλη, το κέρδος που μπορεί να έχουμε από αυτές τις τεχνολογίες. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό ε, κενό, γιατί μπορούμε να μιλήσουμε για τον αντίκτυπο σου σχέση, γιατί ξέρουμε μάλλον την κατάσταση σήμερα στην αγροεργασία, αλλά δεν έχουμε ιδέα για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον και τα πιθανά ωφέλη από αυτέ τι τεχνολογίε. Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα απεσιόδοξοι, να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, αλλά να μην μα τρομάζουν νέε τεχνολογίε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που καταλήγεται σε αυτή την ευχάριστη νότα, γιατί μέχρι τώρα ήταν αρκετά δυσίωνα τα μηνύματα. Αλλά τώρα που ζεσταθήκαμε, νομίζω ότι πιο εύκολα μπορούμε να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες και να αναπτύξουμε τα σχέδιά μας. Όχι τις φαντασιώσεις μας για το μέλλον, αλλά τα σχέδιά μας. Θα δώσω τώρα το λόγο στον δεύτερο αντιπρόεδρο ε, για να προεδρεύσει για το υπόλοιπο της ε, συνεδρίασης. Εγώ από πλευράς μου να σας ευχαριστήσω. Ο κύριος Γολάν τώρα θα προεδρεύσει ε, για το τελευταίο σημείο της μέσης διάταξης για την κοινωνική προστασία των εργαζομένων στην οικονομία πλατφόρμας. Ωραία, προτείνω να αρχίσουμε απευθεία ε, για να δώσουμε έτσι μια συνέχεια στα όσα συζητήθηκαν προηγουμένω. Και βεβαίω έχουμε να κάνουμε εδώ με την κοινωνική προστασία των εργαζομένων στην οικονομία πλατφόρμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά σημαντικό Ω Επιτροπή απασχόληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλαμε και ζητήσαμε να γίνει μια μελέτη σε αυτό το ε, τομέα. Είναι μια σημαντική μελέτη και με περίπου 50 συνεντεύξεις εμπειρογνωμόνων, και στο πλαίσιο της ε, αγοράς αυτής. Ε, νομίζω ότι είναι μια καλή αφετηρία για να έχουμε ορισμένες ε, συστάσεις σε ό,τι αφορά τον τομέα της κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται ραγδαία. Προτείνω να δώσουμε απευθεία το λόγο στους συντάκτες της μελέτης. Έχετε 10 λεπτά έκαστος. Πρώτος ο κύριος Κρίστοφερ Φόρντ και μετά ο κύριος Μάρκ Στιούαρτ. Παρακαλώ κύριε Φόρντ, έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που ε, μας δίνει δυνατότητα να παρουσιάσουμε σήμερα αυτή τη μελέτη η οποία ανετέθη για να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι συνθήκες ε, όσων απασχολούνται στην οικονομία πλατφόρμας. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη μορφή εργασίας. Ε, διότι προσφέρει νέες δυνατότητες ε, για τους εργαζόμενους, ε, περισσότερες ευκαιρίες για ευελιξία. Ο συνάδελφός μας εδώ ανέφερε ότι υπάρχει ένα δυναμικό και για νέες θέσεις απασχόλησης. Πέρα από αυτό υπάρχουν και ερωτήματα που αφορούν για την κατάσταση των εργαζομένων στην οικονομία πλατφόρμας, κυρίως όσον αφορά την νομική τους θέση, ε, κατά πόσον απασχολούνται ως μισθωτοί ε, ή ως ε, ελεύθεροι επαγγελματίες. Και γίνονται και πάρα πολλές συζητήσεις για το κατά πόσον αυτοί οι εργαζόμενοι καλύπτονται από συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή λοιπόν η μελέτη έγινε για να γίνουν όλα αυτά κατανοητά. Ο συνάδελφος Μαρκ Στιούαρτ και Σάμον Τζόις μαζί με μια ομάδα έξι άλλων συναδέλφων ασχοληθήκαμε με τη μελέτη αυτή από το, στο Πανεπιστήμιο του Λίτ. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι το θέμα της κοινωνικής απασχόλησης αντιμετωπίζεται σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν πρόσφατα ενέκρινε μία πρόταση σύσταση προς το Συμβούλιο για προστασία κοινωνική των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων και στόχος είναι οι αποτελεσματικά προγράμματα κοινωνικής απασχόλησης. Υπάρχει και σχέδιο οδηγίας για διαφανείς ε, θέσεις ε, ε, προϋποθέσεις και κριτήρια απασχόλησης. Αυτό αφορά κυρίως τους εργαζόμενους με επισπαλείς συμβάσεις, πολλούς εργαζόμενους της οικονομίας πλατφόρμας. Στόχος της μελέτης είναι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε περισσότερο για το πώς ακριβώς εμπλέκεται η οικονομία πλατφόρμα σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια χρόνια. Πολλές εικασίες ε, υπάρχουν ε, ορολογία για τις μορφές απασχόλησης. Θα εξετάσουμε ορισμένα από αυτά τα θέματα, όπως επίσης και τα κίνητρα της ανάπτυξης στην ε, οικονομία πλατφόρμα. Σημασία έχει να κατανοήσουμε τα ωφέλη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και κάποιες παρενέργειες που προκύπτουν στο θέμα κυρίως της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή η έρευνα ε, έγινε για την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων το 2017. Ε, προβήκαμε σε εντελεχή μελέτη της ε, βιβλιογραφίας και έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα για τους εργαζόμενους οικονομία πλατφόρμας σε πάρα πολλά crowdworking sites. crowd workers και micro workers. Ε, αυτά είναι τα θέματα που εξετάσαμε και πήραμε πάρα πολλές απαντήσεις από αυτού. Κάναμε και αρκετές ε, συνεντεύξεις με άμεσα εμπλεκόμενους σε οκτώ κράτη-μέλη, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ισπανία, Γαλλία, ε, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά τα κράτη-μέλη, ε, σε αυτά ρωτήσαμε εκπροσώπους συνδικάτων, εργαζομένους, ε, πολλούς που εργάζονται σε οικονομία πλατφόρμας, όπως επίσης και όσους χαράσουν πολιτική και διάφορους άλλους που απασχολούνται και εμπλέκονται στην αγορά εργασίας. Ε, πριν σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα, θα ήθελα να γίνει λίγο πιο κατανοητό, ε, να γίνουν κατανοητοί οι όροι που χρησιμοποίησαμε στη μελέτη. Πολλοί όροι χρησιμοποιήθηκαν για να κατανοήσουμε όπως ε, οι επικαλυπτόμενες μορφές απασχόλησης. Στην οικονομία αυτή ακούμε πολύ συχνά για τη συνεργατική οικονομία την οικονομία της μερικής απασχόλησης, sharing economy. Αυτοί είναι ε, όροι, οι δύο πρώτοι χρησιμοποιούνται θετικά για να γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις ε, αυτής της μορφής απασχόλησης, ενώ η επισφαλής gig economy, όπως λέγεται, η ε, περιστασιακή απασχόληση έγινε για να γίνει κατανοητή η επισφαλής απασχόληση. Όλα αυτά αφορούν στην οικονομία πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, περιλαμβάνουμε και την εργασία μετά από αίτημα ε, τα Uber, ε, τους οδηγούς φορτηγών, ε, περιλαμβάνουμε και crowd work όπως είναι η Amazon παραδείγματος χάρη. Δεν συμπεριλάβαμε θέματα που έχουν σχέση με τα Airbnb, τέτοιου είδου site. Όμως τελικά ασχοληθήκαμε με πάρα πολλά που αφορούν στην οικονομία μετά από αίτημα και crowd economy. Αν δει κανείς την βιβλιογραφία θα καταλήξει στο ότι περίπου μέχρι το 5% 1-5% ε, γενικώ ανά τον κόσμο ε, κερδίζουν χρήματα από την οικονομία πλατφόρμας. Ε. Η πραγματική sharing οικονομία δηλαδή ε, τα open source software, ε, το να δανείσει κανείς κάποια αγαθά. Εκεί το ποσοστό όσων προσπορίζονται χρήματα από αυτήν την οικονομία, την οικονομία sharing, ε, είναι πολύ μικρότερο. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η μορφή οικονομίας αναπτύσσεται όλο και περισσότερο και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Εδώ βλέπετε κάποιες ιστοσελίδες, ε, το ένα, μία ιστοσελίδα αφορά τα απορίσματά μας. Και εδώ προσπαθούμε να προβάλλουμε ε, μία έρευνα σε 12.000 εργαζόμενους. Ε, τα πρώτα δύο εδάφια βλέπετε τα πιο σημαντικά ωφέλη ε, που αναφέρουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι ως πλεονέκτημα εφόσον απασχολεί σε αυτή τη μορφή οικονομίας. Για αυτούς λοιπόν ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα να προσποριστούν επιπρόσθετο εισόδημα σε αυτό που έχουν έτσι και αλλιώς. Άλλοι πάλι είπαν ότι έχουν δυνατότητα να εργάζονται από το σπίτι τους. Αυτό αφορά κάποιες μορφές εργασίας, όχι όλες. Αυτούς δηλαδή που χρησιμοποιούν ε, τα click sites, ε, τις ιστοσελίδες αυτές, αυτοί προτιμούν επιθυμούν να εργάζονται το σπίτι και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Επιπλέον όσοι μας απάντησαν μιλάνε και για το ευέλικτο ωράριο εργασίας και αυτό μοιάζει να είναι ένα πολύ βασικό πλεονέκτημα σε αυτές τις μορφές απασχόλησης. Τα επόμενα δύο εδάφια αφορούν στα προβλήματα που μπορούν ε, να προκύψουν. Ε, προσπαθούμε να δούμε πόσο ευχαριστημένοι είναι οι άνθρωποι και προέκυψε το εξής. Πολύ χαμηλή ικανοποίηση όσον αφορά τα επίπεδα ανταμοιβή. Βεβαίω ε, ποικίλει ο χρόνος ε, που δαπανούν οι άνθρωποι ε, στην αμοιβόμενη εργασία και στην οικονομία πλατφόρμας. Είδαμε ότι πολλές φορές στην οικονομία πλατφόρμας είναι χαμηλή η μισθή, άρα δηλαδή η οικονομία πλατφόρμας είναι συμπληρωματική. Επίσης διαπιστώσαμε ότι μόνο ένα τέταρτο από τις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 τους 1.200 εργαζόμενους ε, είπαν ότι είναι ε, πραγματικά ικανοποιημένοι με την ε, αποζημίωση και ακόμα λιγότερο είπαν ότι είναι ικανοποιημένοι με τις ευκαιρίες για να σφυριλατήσουν στα διοδρομία στην οικονομία πλατφόρμας. Κάτι άλλο που βρήκαμε είναι ότι πολλοί χρησιμοποιούν αυτή την μορφή απασχόλησης για συμπλήρωμα. Το 1 τέταρτο όσων απάντησαν είπαν ότι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτή την οικονομία, από αυτή τη δουλειά, δηλαδή, δηλαδή πάνω από μισά από τα εισοδήματά τους τα προσπορίζονται από αυτή τη μορφή της οικονομίας. Ε, χρησιμοποιούμε μία τεχνική Latin Class ανάλυση. Ε, προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε όσους απάντησαν σε διάφορες κατηγορίες χρησιμοποιώντας διάφορες μεταβλητές. Και καταλήξαμε σε τρεις μορφές εργαζομένων σε οικονομία πλατφόρμας με βάση αυτή την ανάλυση. Έχουμε αυτούς που είναι οι μετριοπαθείς εποφελούμενοι, περισσότεροι έχουν λυθεί κάποια άλλη δουλειά. Ε, τα τρία τέταρτα είναι οι σύγχρονοι ε, αποδέκτες, ε, έχουν μεγαλύτερη εξάρτηση από την οικονομία πλατφόρμας. Οι λιγότεροι από τους μισούς κερδίζουν το εισόδημά τους από την οικονομία πλατφόρμας, αλλά αρκετοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες, περίπου το 1 τρίτο είπαν ότι αγωνίζονται ε, κάθε μήνα να τα φέρουν βόλτα. Και μετά υπάρχουν τυχές έρευνες, αλλά καταλήξαμε ότι το 95% έχουν άλλη δουλειά πέρα από την οικονομία πλατφόρμας και φαίνεται ότι δεν εξαρτώνται και πάρα πολύ από την οικονομία πλατφόρμας. Έτσι το 5%, το 50% εξαρτώνται από αυτήν την οικονομία. Βέβαια, ένα μεγάλο ποσοστό, το 27% αντιμετωπίζει κάποιε δυσκολίε από την εργασία πλατφόρμα. Και έχουμε εκείνου που εξαρτώνται πάρα πολύ από την οικονομία πλατφόρμα, Αρκετοί από αυτού, μάλλον λίγοι από αυτού έχουν άλλη δουλειά, εξαρτώνται πλήρω από αυτή τη δουλειά ε, και ε, αρκετοί έχουν πάνω από το μισό εισόδημά τους από αυτήν την μορφή εργασίας και πολλοί έχουν δυσκολίε να τα φέρουν βόλτα. Για να ολοκληρώσω θα ήθελα να επισημάνω κάποιες ε, προκλήσεις. Ε, σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη επισφάλεια όσον αφορά αυτή τη μορφή εργασίας. Και αυτό σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα ένα κομμάτι αυτών των εργαζομένων εξαρτώνται απόλυτα από αυτή τη μορφή εργασίας για το εισόδημά τους. Υπάρχουν κάποιοι εργαζόμενοι που δεν έχουν κοινωνική προστασία, άρα δηλαδή όσο περισσότερο εξαρτώνται από αυτή τη μορφή εργασίας, τόσο λιγότερη κοινωνική προστασία απολαμβάνουν. Και αυτό το βλέπουμε με διάφορους τρόπους. Πρώτα απ' όλα ε, η θέση τους, η απασχόληση. Έχουν ανεξάρτητες συμβάσεις, δηλαδή εξαιρούνται πλήρως από οποιαδήποτε μορφή κοινωνικής προστασίας και επιπλέον εξαρτούνται, ε, αποκλείονται μάλλον, με αποκλείονται και από ε, τα ωράρια εργασίας που έχουν καθιερωθεί. Το δεύτερο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι ενώ η προστασία υπάρχει για εργαζόμενους, η κοινωνική προστασία, αυτή όμως ε, προκύπτει για μορφές απασχόλησης εκτός της οικονομίας πλατφόρμας, από στάνταρτ μορφές απασχόλησης ή από τα δικαιώματά τους ως πολίτες. Αυτό προϋποθέτει η πύλη προς την κοινωνική απασχόληση προκύπτει από τις κλασικές μορφές απασχόλησης και όχι τόσο από τις άτυπες ε, μορφές απασχόλησης όπως είναι η εργασία σε οικονομία πλατφόρμας. Η άλλη δουλειά που έχουν οι περισσότεροι στην κλασική οικονομία και αυτή όμως είναι αρκετά επισφαλής, Άρα δηλαδή, ενώ κάποιοι από αυτούς τους εργαζόμενους έχουν κάποια προστασία από άλλες ε, θέσεις απασχόλησης και αυτή η άλλη μορφή απασχόληση είναι ε, παροδική, είναι επισφαλής, άρα αυτή είναι διπλά επισφαλής και στην οικονομία πλατφόρμας και στην κλασική οικονομία. Και ως εκ τούτου προκύπτουν αρκετές προκλήσεις για την κοινωνική προστασία. Αυτή τη στιγμή εμείς ε, θέλουμε να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση ε, αλλά υπάρχουν αρκετές ε, προκλήσεις για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι μορφές απασχόλησης θα περιλαμβάνονται στην κοινωνική απασχόληση. Πρέπει να υπάρξει κάποια αναθεώρηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης να περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι στην ε, οικονομία πλατφόρμας. Το ελάχιστο εισόδημα, αυτό είναι πρόβλημα για κάποιους εργαζόμενους, δεν φτάνουν σε αυτό το ελάχιστο εισόδημα για να μπορούν να απολάβουν κοινωνικών δικαιωμάτων. Εξάλλου, όταν αυτοί ε, μετακινούνται από μία θέση απασχόλησης πλατφόρμα σε άλλη, δεν εποφελούνται από κοινωνικές μορφές προστασίας. Εξάλλου προτείνουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια θεμελιώδη δικαιώματα για όλες αυτές τις μορφές απασχόλησης, για όλους τους πολίτες. Αυτό θα ήταν μια επικοδομητική πρωτοβουλία. Δηλαδή οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες και όσοι δεν επωφελούνται απο κοινωνικες μορφες προστασιας εξαλλου προτεινουμε οτι θα πρεπει να υπαρχουν καποια θεμελιωδη δικαιωματα για ολες αυτες τις μορφες απασχολησης αυτό το καθεστώς, αυτοί θα πρέπει να μπορούν να απολάβουν ε, κάποια βασικά δικαιώματα. Ε, στη μελέτη μας διαπιστώσαμε επίσης ε, ότι υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες, τα βασικά δικαιώματα για πολλούς σημαίνουν κοινωνική προστασία που θα συμπληρώνεται σε εθνικό επίπεδο από σχετικούς κανονισμούς και σχετική νομοθεσία. Και το τελευταίο που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι εθνική εθνικές στατιστικές υπηρεσίες θα πρέπει να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για αυτή τη μορφή απασχόλησης, αλλά και να ε, θέσουν σε εφαρμογή διαδικασίες ε, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν δεδομένα για, την, το εύρος, την έκταση στην οποία ε, εργάζονται αυτοί οι απασχολούμενοι υπάρχει η δυνατότητα οι εργαζόμενοι αυτοί να εκπροσωπούνται μέσα από συνδικάτα, από, ε, από ενδιάμεσους στο χώρο εργασίας. Ε, βεβαίως διαφέρουν πάρα πολύ τα δεδομένα αναχώρα ε, σχετικά με το κατά πόσο αυτές οι νέες μορφές απασχόλησης μπορούν πραγματικά να καταλήξουν και σε ουσιαστική εκπροσώπησή τους. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε τη δυνατότητα να να σας παρουσιάσουμε σήμερα την εργασία μας και βεβαίως με μεγάλη μας χαρά. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση, ευχαριστώ για την εκθεσή σας. Πρέπει να πω ότι μιλώ εκ μέρους και του συναδέλφου, ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα της εργασίας σε πλατφόρμες Και αυτό το οποίο μας ικανοποιεί για τη μελέτη ε, είναι ότι όπως οι πολλοί... Και για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, ε, σίγουρα είναι σημαντική η συμβολή σας. την Επιτροπή η έλλειψη δεδομένων. σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μας λένε ότι δεν ξέρουμε ε, περί τίνος πρόκειται και δεν ξέρουμε αν πρέπει να λάβουμε μέτρα. Επομένως μας βοηθάτε να συμπληρώσουμε αυτό το κενό για την εξέλιξη των ε, πολιτικών. Ότι αφενός η μελέτη καταδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχει πολιτική, δράση από πλευράς πολιτικής για να διαμορφώσουμε την εξέλιξη της οικονομίας πλατφόρμας ε, με δίκαιο και βιώσιμο τρόπο από κοινωνική σκοπιάς και πόσο περίπλοκες ε, είναι οι διάφορες πλατφόρμες. Γιατί ναι, μεν υπάρχει μια ποικιλομορφία, αλλά ποικιλομορφία υπάρχει και στο επιχειρηματικό τοπίο, ε, στην ε, παραδοσιακή οικονομία. Υπάρχουν ομοιότητες και αυτή η μελέτη μας βοηθά να τις μελετήσουμε. Ο ρυθμιστικός στόχος, ήρθε και ο γειτονά μου εδώ, καλωσορίσατε, δικτύου. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουμε εμείς και πρέπει να υπάρχουν τα ίδια δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις για όλους. δεν θα πρέπει οι επιχειρήσεις της οικονομίας πλατφόρμας να μπορούν να ελαχιστοποιήσουν ε, τις υποχρεώσεις τους και να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επειδή παρακάμψια για να δούμε τι ε, πραγματικά το υπάρχει σε επίπεδο εργασίας και να φροντίσουμε η νέα, εργασία, ε, η νέα νομοθεσία να είναι χωρίς αποκλεισμούς και να περιλαμβάνει όλες τις νέες ευέλικτες μορφές εργασίας. Ωστόσο, πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπέρα και ζητούμε μια ευρωπαϊκή αρχή στην οικονομία πλατφόρμας. Μια πρόσφατη μελέτη ε, η οποία απασχόλησε τον συνάδελφο είναι μια μελέτη του Φρίντριχ Έμπερχαρτ Σίφτον η οποία δείχνει ότι η ευρωπαϊκή προσέγγιση ε, είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο οδηγία για την ε, εργασία σε πλατφόρμα και η μελέτη φαίνεται να έχει και κάποιες επιφυλάξεις και να μην ζητά συγκεκριμένη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια παραπάνω πράγματα γι' αυτό. Δεύτερον, ε, ταξινόμηση των εργασιακών σχέσεων βάσει προσόντων. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοαπασχολούμενοι. Όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, ε, ότι το βάρος της απόδειξης ε, επαφίεται στον εργαζόμενο αν θέλει να αποδείξει ότι είναι κάτι άλλο και είναι και η πιο αδύναμη σε αυτή την ε, εργασιακή σχέση κατά πάσα πιθανότητα. Επομένως, μία πιθανή λύση σε αυτό το πρόβλημα η σχέση για την παροχή εργασίας πλατφόρμας είναι μία σχέση απασχόλησης μεταξύ του εργαζομένου στην πλατφόρμα και της πλατφόρμας. Να μην βαρύνεται δηλαδή ο εργαζόμενος αλλά η πλατφόρμα και εν τέλει να είναι μόνο, υπησέρχονται όλες οι διάφορες δυνατότητες. Μόνο η πλατφόρμα μπορεί να δώσει πραγματικές αποδείξεις για την πραγματική σχέση που υπάρχει. Και αυτή η νομική υπόθεση ισορροπίας που υπάρχει και τη δυνατότητα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες. Η ερώτησή μου είναι κατά πόσον θεωρείτε ότι είναι εφικτή αυτή η λύση και κατά πόσον το έχετε συζητήσει στα πλαίσια αυτής της μελέτης και κάτι πιο γενικό, είπα σωστά, για το πώς θα βελτιωθεί η κοινωνική κατάσταση των εργαζομένων στην οικονομία πλατφόρμας και αν μπορούμε ε, να το κάνουμε αυτό χωρίς να αλλάξει το βάρος της απόδειξης. Βάσει των αυτοαποσχολούμενων και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση. Λοιπόν, να ξεκινήσω και μετά θα το τι συζητήσαμε ως ερευνητές όταν γράφαμε την έκθεση. Ε, έγιναν πολλές συζητήσεις για κάποια από αυτά που μόλις αναφέρετε, για την ε, νομική ταξινόμηση, κατάταξη ε, και τις πιθανές απαντήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νομικός εμπειρογνώμονας μας δεν είναι εδώ